Να ξεκινήσουμε. Καθίστε παρακαλώ. Έχουμε καθυστερήσει και λίγο. Είναι 10 και 8 λεπτά, αν βλέπω καλά. Παρακαλώ καθίστε για να ξεκινήσουμε. Και στην αρχή θα ήθελα παρακαλώ να σας ζητήσω να φορέσετε τα ακουστικά σας για να ακούσετε ένα σύντομο μήνυμα από τους διερμηνείς μας. Οι διερμηνείς θα ήθελαν να μας πούν δύο λόγια. Παρακαλώ, πριν την ψηφοφορία, φορέστε τα ακουστικά σας. Φορέστε τα ακουστικά σας παρακαλώ για να ακούσετε το μήνυμα των διερμηνέων. Βρισκόμαστε στην τρίτη εβδομάδα κινητοποιήσεων λόγω τη εργασιακή διένεξη με τη διοίκηση για τι συνθήκε εργασία μα. Σε ορισμένε καμπίνε έχουν επιστρατευτεί όλοι οι διερμηνεί και είναι υποχρεωμένοι να εργαστούν.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 Δεν μπορούμε να παρατείνουμε την, την συνεδρίαση πέραν της 12.30 γιατί δεν θα έχουμε διερμηνία μετά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, για την ανακοίνωση και περνάμε στην ψηφοφορία. Ας κάνουμε πρώτα έναν έλεγχο των μηχανημάτων. Δοκιμαστική ψηφοφορία, λοιπόν. Άρχεται η ψηφοφορία. Παρακαλώ, ψηφίστε για να ελέγξουμε το μηχάνημα. Τέλος ψηφοφορίας. Νομίζω ότι το μηχάνημα λειτουργεί. Και να περάσουμε στις ψηφοφορίες. Το πρώτο θέμα προς ψήφιση αφορά τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Βιομηχανικής Ανάπτυξης του τομέα της άμυνας. Η συγγήτρια είναι η κυρία Γκροστέτ. Θα ψηφίσουμε την προσωρινή συμφωνία μετά τον άτυπο τριμερή διάλογο. Θα γίνει η ψηφοφορία με ονομαστική κλίση και κυρίσω την έναρξη της ψηφοφορίας. Τέλος ψηφοφορίας. Ένας υπεράριθμος από το ΕΛΚ έχει παρατηρηθεί. Εντάξει, εντάξει τώρα, ωραία, τέλεια. Τέλος ψηφοφορίας. 47 ψήφοι υπέρ, άρα γίνεται δεκτή η προσωρινή συμφωνή και συγχαρητήρια στην εισηγήτριά μας, την κυρία Γκροστέτ, για το αποτέλεσμα. Προχωράμε στο σημείο 10 την Ευρωπαϊκή Κοινή Επιχείρηση Πληροφορικής Υψηλών Επιδόσεων. Ο εισηγητής μας είναι ο κύριος Σιγμάντας μπαλτσίτη. Ψηφίζουμε την τροπολογία 65. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 66 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 67 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 88 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 89 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 97 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται από ό,τι καταλαβαίνω. Παρακαλώ να σηκώνετε καλά τα χέρια σας. Τροπολογία 98 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 4α, συμβαστική 4α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 12 υπέρ κατά απόχέ, εγκρίνεται. Τροπολογία 107 υπέρ κατά Ηλεκτρονικό έλεγχο παρακαλώ και την τροπολογία 107 άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Πάλι έχουμε έναν υπεράριθμο από το ΕΛΚ. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 108 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 109 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 110 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 110. Άρχεται η ψηφοφορία. Και πάλι έχουμε έναν υπεράριθμο από το ΕΛΚ. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 114 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 115 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 116 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 117 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 119 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 120 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 121 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 122 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 123 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 124 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 125 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 126 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 127 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 128 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 129 υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος για την 129 άρχεται η ψηφοφορία Τέλος. Απορρίπτεται. Τροπολογία 130. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 135 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 15 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 26 υπέρ κατά αποχές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 αποχές απορρίπτεται. 52 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 53 υπέρ. Κατά αποχές και ο ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 53. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 60 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 62 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία μετά τις τροπολογίες με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Και εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον εισηγητή μας, τον κύριο Μπαλτσίτης. The next. Πάμε τώρα στην επόμενη ψηφοφορία που είναι το σημείο παριθμών 11. Πρόθεση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών. Κλωτούρμες, ο εισηγητής μας. Που παρίσταται για τελευταία φορά στην Επιτροπή. Αλλά και η κυρία Κάλλας για τελευταία φορά είναι μαζί μας. Ξέρετε, από την αρχή της θητείας πριν από τέσσερα χρόνια δηλαδή, ο Σίτρα, 11 συνάδελφοι πήγαν στις κυβερνήσεις των χωρών τους ως υπουργοί. Να, Βγάζει υπουργού η Επιτροπή και μην το ξεχνάτε. Αν θέλετε να γίνετε υπουργό, τη γνώση τη χώρα σα, θα πρέπει να κάτσετε εδώ. Εδώ, στην επόμενη θητεία. Στα σίγουρα στο λέω. Τέτοιε επιδόσει δεν έχει καμία άλλη επιτροπή. Να το θυμάστε. Και δεν λέω για πρωθυπουργό, είναι αυτό είναι άλλο θέμα. Εκεί όλοι έχουμε πιθανότητα. Μην το ξεχνάτε. Βλέπω, συμφωνείτε μαζί. Πολύ ωραία. Πρώτη καθαρά από δικών οχημάτων οδικών μεταφορών. Κλώτσε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνεργασία. Και εσένα, καλή. Wow, wow. Θα τα λέτε στο Συμβούλιο και φαντάζομαι θα υποστηρίζετε εμά και όχι το Συμβούλιο. Να μας θυμάστε. Πολύ ωραία. Επομένως, τον 32, 17, 18 και το 29. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται προφορική τροπολογία. Υπάρχουν ενστάσεις. Επομένως, υπέρ. Εμείς έχουμε ένσταση. Πόσοι. Αν έχουμε πάνω από τέσσερις. Πόσοι είστε. Τρεις ή τέσσερις. Παρακαλώ. Σηκωθείτε εσείς που ενίσταστε. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ. Οπότε δεν θα γίνει η ψηφοφορία. 30. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 81. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Περνάει. Και εγκρίνεται. Επόμενη. Δεν βλέπω τι ψηφίσατε. Το 82 και το 84. Πέρασε ψηφοφορίας. Και απορρίπτεται. 31 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 83 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 85 88, 94, 101, 103, 142, υπέρ, κατά, έλεγχος για όλες αυτές και οι έξι αυτές τροπολογίες. Ψηφίζουμε, πέρας. Εγκρίνεται. 36. Αν εγκρίνεται πάμε στο Στη σελίδα 6, σελίδα 6. Για την 36. Σας περιμένω. 36. Μήπως είναι στο 5. Συμπαθάτε με, γιατί έχω άλλη εκδοχή το κείμενο. Έτοιμοι. Ναι, ωραία. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 106 υπέρ έλεγχος για το 36 καλώς ίσως δεν ήσασταν έτοιμοι να ψηφίσετε ο κατάλογος δεν απορρίπτεται πέρα ψηφορίας απορρίπτεται 106 υπέρ κατά έλεγχος για το 106 Πέρας. Απορρίπτεται. 107 υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Παρακαλώ, σηκώστε το χέρι σας με τρόπο να είναι εμφανές. Είναι εμφανές τι ψηφίζετε πέρα ψηφορίας και απορρίπτεται. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά έλεγχος για την πρώτη συμβαστική. Πέρασε. Εγκρίνεται. Και πάμε στο 37. 108, 109, 110 και 111. Όλες μαζί υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. «115, 119, 149 και 154 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 122 στη σελίδα 10 στο δική μου εκδοχή του κειμένου. 122 επαναλαμβάνει ο πρόεδρος. Ανάτι. 122. Του βρήκατε. Ωραία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. απορρίπτωται. Η 38 αποσύρεται. 123 υπέρ. Κατά. Ας γίνει ηλεκτρονικός έλεγχος καλύτερα. 123 έλεγχος. Πέρας εφορίας. Rejected. 39 and 26 in favor. Against Abstention rejected. Απορρίπτεται. Η επόμενη είναι 124 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται 125, 73 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. Οι 40 και 27 αποσύρονται. 126 υπέρ κατά έλεγχος. 126. Πέρασε ο φορείας. Απορρίπτεται. 127, 128 και 76 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 41 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 129 και 71 υπέρ κατά έλεγχος. Voting. And I close the vote. One EPP too many. Uh, one EPP too many. One... Πάλι ψήφισε ένας παραπάνω από το έλεγχο όμως. I close the vote. Πέρασε. Και απορρίπτωται. 130 in favor. 130 υπέρ. Κατά, ας γίνει έλεγχος για να ξέρουμε ακριβώς το αποτέλεσμα. 130. Πέρασε. Εγκρίνεται. 131 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά. απορρίπτεται με σαφή πλειοψηφία. 42 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σε τι ψηφίζεται. Δεν σηκώνετε κατά 42 λέω. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 132 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 3. Υπέρ κατά έλεγχος για την τροπολογία 3. Πέρασε οφορίας. Απορρίπτεται. 49 υπέρ. Κατά. Και πάλι ηλεκτρονικός έλεγχος για το 49. Απορρίπτεται. 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 6 Παρακαλώ συνάδελφοι, παρακολουθείτε την ψηφορία. 5 και πάλι. Το 5 Δεν βλέπω τι ψηφίζεται. Πέρα και απορρίπτονται. 6. 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 53. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Για το 53. Πέρα εγκρίνεται αυτή τη φορά. Επτά. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Για το επτά. Πέρασε ο Απορρίπτεται. Οκτώ. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Πέρα τη ψηφοφορίας. Εννέα, υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. Την ίδια πλειοψηφία. 10, υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 11 υπέρ κατά έλεγχος. 11. 11 πέρα ψηφοφορίας. Με ευρία πλειοψηφία εγκρίνεται 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 61 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16 υπέρ κατά απορρίπτεται 65 υπέρ κατά αποχές το 63 υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Για το 36. 63, 63 διορθώνει. 63 διορθώνει. 63, I close the vote. Πέρασε τη οφορία. το 63. 62 υπέρ. Κατά. Αποχές έλεγχος. Πέρα της εφορία. Εγκρίνεται 64, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 68, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 69, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται 70, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 23. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος για τη συμβαστική 4. Παρακαλώ να σηκώνετε εμφανώς το χέρι. 4. Πέρα ψηφοφορίας. Ναι, εγκρίνεται όπως ε, είπαμε 23 υπέρ. Κατά. εκεί, έλεγχος για το 23. Έλεγχος. Πέρας. Απολύτως. 24 υπέρ. Κατά. Έλεγχος. 24 πέρα της εφορία. Απορρίπτεται 25 υπέρ. Κατά. Και πάλι ένοχο. Πέρα εφορία. Απορρίπτεται. Το 25 και πάμε στο 28 υπέρ. Κατά. Το 28. Πέρασε ο φορείος. Απορρίπτεται. 78. Χωριστή ψηφορία, Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Είμαστε διχασμένοι από γίνει έλεγχος για το πρώτο τμήμα. Πέρα σοβαρίας. Πενήντα. Εννέα. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Πέρα σοβαρίας. Απορρίπτεται. 80 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τελική ψηφοφορία, ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Ονομαστική ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται to draft report, which is uh, point of order, Mr. Υπάρχει ένα διαδικαστικό, κύριε Πρόεδρε, λέει ο γραμματέα από τον κύριο Τούρμες. Θα ήθελα να αποσύρω την ε, υπογραφή μου την έκθεση. Απορρίφθηκε τώρα η έκθεση και νομίζω ότι τα επόμενα φεντικά στην Ευρώπη θα πρέπει να λάβουν υπόψη τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα λεωφορεία, τα λεωφορεία, συγγνώμη. Θα πρέπει να λάβουμε πλέον καθαρή ενέργεια, υδρογόνο κλπ. Δεν ξέρω, ίσως έχασα τη, μαγεία στην επιρροή μου. Οπότε δεν ξέρω, μήπω γι' αυτό πια πρέπει να φύγω. Τέλος πάντων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέρασα πολύ ωραία. Ε, thank ε, Εμείς ευχαριστούμε κύριε Τούρμες, λέει ο πρόεδρος. Ευχαριστούμε Κλοντ. Προχωρούμε τώρα στο σχέδιο έκθεσης που αφορά έναν κανονισμό. Κατάργηση του κανονισμού 256 του 14 και αφορά τα πνευματικά σχέδια σε ενεργειακή υποδομή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συγκέντρια είναι η κυρία Μπαρμπαρα θα ψηφίσουμε μαζί για αρχή τις τροπολογίες 1 και 2 υπέρ κατά ζητείτε ονομαστική ψηφοφορία. Καλά, ό,τι θέλετε. Έχετε δίκιο, λέει ο Πρόεδρος και συμπαθάτε με. Γιατί πρόκειται για απόρριψη της ε, πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οπότε θα γίνει ονομαστική ψηφοφορία πέρα ψηφοφορίας. και απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία. Η ονομαστική ψηφοφορία επίσης ψηφίζουμε. Πέρασε ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια. Στην εισηγήτρια και τώρα πάμε στο επόμενο και έκθεση. Πρώτη για την πρώτη ε, τροποποίηση του Μνημονίου Συνεργασίας Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγχαρητήρια είναι ο Ρολάντας Πάξας. Με ηλεκτρονικό τρόπο θα κάνουμε ονομαστική ψηφοφορία και ψηφίζουμε. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε πέρα ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και σας ευχαριστώ συνάδελφοι. Και η επόμενη έκθεση είναι του Ρολαντάς Πάξας και έχουμε την παράταση της συμφωνίας για επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Πέρα ψηφοφορίας. Το ίδιο αποτέλεσμα. Συγχαρητήρια. Πάμε τώρα στην τελευταία μας ψηφοφορία. Συμφωνία Συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και Οργανισμού για Ασφάλεια Αεροναυτιλίας στην Αφρική και Μαδαγασκάρη. Ο υποφαινόμενος είναι ο συγητής, ψηφίζουμε. Πέρα ψηφοφορίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Τελειώσαμε τις ε, ψηφοφορίες και σας ευχαριστώ συνάδελφοι. Παρακαλώ μην ξεχνάτε ότι έχουμε ακόμα πολλή δουλειά και θα πρέπει να ολοκληρώσουμε τις ε, εκθέσεις πριν τις 10 Ιουλίου. 10 Ιουλίου. Όλες τις εκθέσεις. Και είναι πολλές. Βέβαια, εξαιρείται που πάει στις 19 Ιουλίου η έκθεση για το πρόγραμμα πλαίσιο. 10 Ιουλίου. Πάρα πολύ σημαντικό και δύσκολο. Okay. Uh, we will go... Και τώρα πάμε στο επόμενο σημείο της σημερινής διάταξης. Σε τρία λεπτά. Μην φύγετε. Κανένας. Good. Ladies and gentlemen, uh, sorry, uh, uh, let me say... λέει ο θα πρέπει να καλωσορίσουμε τον κύριο Ντομινίκ Ριστορή. Είσαστε μονίμως προσκεκλημένος του Κοινοβουλίου. Άρα τίποτα το εξαιρετικό και το περίεργο που ήρθατε, γιατί έχουμε το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη που αφορά το μηχανισμό συνδέοντας την Ευρώπη και έχουμε τώρα κάποια είδους ε, ε, ενημέρωση για τις ε, διαπραγματεύσεις. Είναι το τελευταίο θέμα που θα συζητήσουμε πριν την μεσημβρινή διακοπή. Και έχουμε τον συνάδελφο Μύροσλαβ Κόχε, ο οποίος θα μας ενημερώσει όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για την αποτελεσματική χρήση της ενέργειας. Δεν ξέρω αν είστε ενημερωμένοι, αλλά σχεδόν έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδρομή του θέματος. Δεν τελειώσαμε το θέμα στη συνάντηση της Ολομέλειας του Στρασβούργου, οπότε το αναβάλαμε. Πάντως, ο Μύρος βρίσκεται εδώ και συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Οπότε, αυτό που θα είναι πιο εξυπηρετικό για εκείνον είναι να μας πει τώρα δύο λόγια όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις. Τώρα, τώρα και όχι σε μία ώρα. Γιατί πρέπει να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις στο Συμβούλιο και να συζητήσει με Συμβούλιο και Επιτροπή όλες τις ε, λεπτομέρειες για να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις πριν τις 7 πριν τις 7 μετά μεσημβρία απόψε. Οπότε και θα αρχίσει η συζήτηση για τη διακυβέρνηση. Άρα θα πρέπει για την απόδοση και αποτελεσματικότητα να ολοκληρωθεί το θέμα πριν τη διακυβέρνηση της Ενδιακής Ένωσης. Επίση, θα πρέπει να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσει για τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια που έχει αναλάβει ο συνάδελφο Μπλάνκο Λόπεθ. και εκείνος έχει ένα θεματάκι που πρέπει να διεκπαιριωθεί. Πάντως, είναι άσχετο, άσχετο το παγκόσμιο κύπελο εν προκειμένου. Μύροσλαβ Πόχε. Μπορείς ε, να μα πει δύο λίγων τι γίνεται σε ένα τριλεπτάκι. Διλεπτάκι, διλεπτάκι. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ε, μου δίνετε εδώ να μιλήσω νωρίτερα. Να σας ενημερώσω πολύ σύντομα σχετικά με το τι συμβαίνει ε, με την ενεργειακή απόδοση. Ε, υπήρξε μια συμφωνία σε τεχνικό επίπεδο και τη χαιρετήσαμε. Συμφωνήσαμε σε όλα τα τεχνικά θέματα και πρέπει να σας πω ότι θα ήθελα να ευχαριστήσω την διαπραγματευτική ομάδα του Κοινοβουλίου αλλά και της Επιτροπής που κατέληξαν σε συμβασμό. Απομένουν τρία θέματα που πρέπει να συζητηθούν. Ε, το επίπεδο των στόχων, άρθρο 7 και άρθρο 3, σχετικά με την ε, πρωτογενή ή την τελική μορφή ενέργειας. 11 Ιουνίου συναντήθηκαν οι Υπουργοί Ενέργειας και οι δύο θεσμοί παρουσίασαν τι θέσει τους. Ήταν πολύ κοντά στο να βρουν έναν αποδεκτό συμβασμό με την Προεδρία αυτά την περασμένη Πέμπτη. Τελικά όμως ε, δεν επιτεύχθηκε συμφωνία παρότι πλησίασαν θέσει θέσεις των δύο θεσμών. Αλλά σας λέω, δεν καταλήξαμε σε συμβιβασμό για να συνδυάσουμε τα τρία πολιτικά θέματα, ε, για να είναι όλα αποδεκτά για τους ε, θεσμούς. Ε, θα υπάρξει λοιπόν ένας άλλος γύρος διαπραγματεύσεων, μόλις μόλις φύγω από εδώ και ελπίζω να καταλήξουμε σε μια συμφωνία έτσι ώστε να υπάρχουν αρκετά υψηλοί στόχοι ε, και ως προς τους στόχους Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και σε σχέση με το άρθρο 7. Ε, θα μπορούσαμε να καταλήξουμε κατά 32,5% όσον αφορά το, τη μη δεσμευτική φύση του στόχου. Και οι δύο θεσμοί είναι έτοιμοι να επιτρέψουν μια νέα αναθεώρηση έτσι ώστε το επίπεδο των στόχων να συμπεριληφθεί στο 2023. Όσον αφορά το άρθρο 7, νομίζω ότι τελικά θα μπορέσουμε να καταλήξουμε στη συμφωνία όσον αφορά το πραγματικό επίπεδο ετήσιας εξοικονόμησης ε, που πρέπει να επιτύχουν τα κράτη-μέλη μετά το 2020. 0,71% είναι το επίπεδο της εξοικονόμησης τώρα και ελπίζω να αυξηθεί, να καταλήξουμε σε ένα συμβασμό από 7,8 μέχρι 0,7 μέχρι 0,7 9%. Ελπίζω λοιπόν ότι με τον τρόπο αυτό θα καταστεί δυνατόν να κλείσουν σήμερα οι διαπραγματεύσει και έτσι θα καταστεί δυνατόν και να κλείσει και όλο αυτό το θέμα. Όπως βλέπετε λοιπόν, υπάρχουν μόνο για σήμερα τρεις τριμεροί διάλογοι. Μόνο για σήμερα διακυβέρνηση, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και απόδοση. Ε, θέλουμε να κλείσουν σήμερα ή δυνατόν και οι τρεις ε, ή το πολύ πολύ αύριο μέχρι τις 5 ε, το πρωί ή 4 το πρωί. Δεν ξέρω. Εμείς, αν θέλετε, δεν έχουμε πρόβλημα να παραμείνουμε μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις και για τα τρία θέματα. Να κλείσουν όμως όλα σήμερα μέχρι αύριο το βράδυ και μέχρι τις 27 Ιουνίου όπου θα ξεκινήσουμε με το σχεδιασμό της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Τις 27 αυτά. Τα επόμενα θέματα θα αφαιθούν στην Αυστριακή Προεδρία. Ελπίζω όλα αυτά να συζητηθούν τον Ιούλιο γιατί ζητήσαμε ε, με τα θέματα αυτά να επιληφθεί η Αυστριακή Προεδρία. Και γιατί είναι τόσο σημαντικά όλα αυτά τα θέματα αγαπητοί συνάδελφοι. Αναφέρομαι συγκεκριμένα στον Άσερ και στην ετοιμότητα για κινδύνους. Αυτά τα δύο θέματα θα εξετάσει η Αυστριακή Προεδρία. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει οι διαπραγματεύσεις να ξεκινήσουν τον Νοέμβρη και έχουμε 12 νομοθετικές προτάσεις ε, για, ε, για διαπραγμάτευση. Αυτό θα ξεκινήσουν αρχές Δεκεμβρίου. Θα ξεκινήσουμε με την Αυστριακή Προεδρία, μετά θα περάσουμε στη ε, Προεδρία της ε, Ρουμανίας. Αυτά τα θέματα της ενέργειας να κλείσουν το συντομότερο δυνατόν. Γιατί αλλιώ δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε να τα καταφέρουμε σχετικά με τον προϋπολογισμό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μύροσλαβ, ε, ευχαριστούμε εσάς και τον ε, συνάδελφό μας, ε, τη συνάδελφό μας, κυρία Λόπες, τον, τον, με συγχωρείτε, τον κύριο Λόπες. Ευχαριστούμε και τον κύριο Τούρμες και όλοι μας ε, θα εργαστούμε πολύ σκληρά για να τελειώσουμε σήμερα και αύριο. Πάμε στο επόμενο θέμα, Connecting Europe Facility, ο μηχανισμός συνδέοντας την Ευρώπη έχουμε τον Γενικό Διευθυντή, τον κύριο Ριστόρη, ο οποίος θα μας παρουσιάσει το θέμα αυτό. Και ο προπλογισμός του 2021-2027, ένα κομμάτι αυτού, εκεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε πρόσφατα να ανανεωθεί αυτός ο μηχανισμός συνδέοντα στην Ευρώπη για να στηρίξουμε τις επενδύσεις ε, στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υποδομών και εμεί ε, θα είμαστε αρμόδιοι για την ενέργεια και τα ψηφιακά, αποκλειστικά αρμόδιοι και εν μέρη αρμόδιοι και για τα θέματα των μεταφορών. Στον τομέα της ενέργειας 8,2 δις ε, προβλέπονται, περίπου 9 δις ευρώ, ε, για να στηρίξουμε επενδύσεις, έτσι ώστε να προαχθεί η ενεργειακή αγορά και η ενεργειακή μετάβραση να συμβαδίζει με τους στόχους της καθαρής ενέργειας, ε, δηλαδή το δικό μας το πακέτο που αναφέραμε πριν από, λίγο, πριν από λίγα λεπτά. Ο Γενικός Διευθυντής προσεκλήθη για να μας παρουσιάσει το ενεργειακό κομμάτι αυτής της πρότασης για την ανανέωση του μηχανισμού συνδέοντας στην Ευρώπη και για να μας παρουσιάσει και λεπτομέρειες αυτού του θέματος. Κύριε Γενικέ, για μας το θέμα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θέλουμε να ενημερωθούμε σχετικά με τα σχέδιά σας, το πώς ακριβώς ε, βλέπετε αυτό το μηχανισμό συνδέω στην Ευρώπη κατά την αμέσως ε, επόμενη περίοδο. Είναι πολύ σημαντικό γιατί θέλουμε, σας είπα, να κλείσουμε το θέμα της ενέργειας και εσείς ε, είσαστε κατά κύριο λόγο αρμόδιος για θέματα ενέργειας, εν μέρη και για θέματα ψηφιακά. Παρακαλώ, Ντομινίκ, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμη Ευρωβουλευτέ, όπως ξέρετε, ε, βαδίζουμε όλο ταχώς προκειμένου να θεσπίσουμε στην Ευρώπη το πιο προηγμένο νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο για την ενέργεια στην Ευρώπη. Με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ιδιαίτερα με την υποστήριξη της Επιτροπής Ήτρε, της δικής σας Επιτροπής. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να μην ξεχνούμε ότι το κανονιστικό πλαίσιο στις ενεργειακές υποδομές θα πρέπει ε, με τις, θα πρέπει να συμβαδίζει με τις υποδομές μάλλον. Ε, είναι αδύνατον να έχουμε εντυπωσιακά αποτελέσματα χωρίς να ε, αντιμετωπίζουμε ταυτόχρονα το ρυθμιστικό πλαίσιο με τις υποδομές. Θα πρέπει το θέμα του νομοθετικού ρυθμιστικού πλαισίου να συμβαδίζει με τις υποδομές. Αυτό ισχύει και για τις προτεραιότητες της ενέργειας, αλλά και για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Θα θυμάστε την ε, κατάσταση που είχαμε ε, πριν από 10 περίπου χρόνια με τη μεγάλη κρίση στην Ουκρανία. Και είναι σημαντικό και στα πλαίσια της διαφοροποίησης ε, το θέμα της ενεργειακής ασφάλειας. Θα πρέπει πρώτα να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις λόγω των τροτών σημείων πολλών χωρών, ιδιαίτερα στην ε, κεντρική, ανατολική αλλά και στην ε, νότιο-δυτική Ευρώπη, δηλαδή και στην ανατολική και στην βόρεια Ευρώπη, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και όλες τις πτυχές της ανταγωνιστικότητας. Μια καλά, ένα καλό ολοκληρωμένο δίκτυο ενισχύει τον ανταγωνισμό, αλλά ταυτόχρονα ε, οδηγεί και σε πιο ανταγωνιστικέ τιμέ, κάτι που είναι επίση πολύ σημαντικό. Το ίδιο όμως ισχύει όλο και περισσότερο ε, στο θέμα της βιωσιμότητα. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την πρόκληση της ολοκλήρωσης, ε, όλο και περισσότερο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Και αυτό ενδιαφέρει τόσο την αγορά όσο και την ασφάλεια του των ευρωπαϊκών δικτύων. Για παράδειγμα, η Πορτογαλία παρήγαγε το Μάρτιο πάνω από 100% ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, χωρίς κοινή διαχείριση του δικτύου με την Ισπανία, αυτό θα είχε δημιουργήσει πολλές δυσκολίες σε ό,τι αφορά τη διαφύλαξη της σταθερότητας του δικτύου. Επίσης, έχοντας κατά νου όλα αυτά τα νευραλγικά θέματα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ένα νέο μηχανισμό συνδέοντας την Ευρώπη με ένα νέο κονδύλιο 8,65 δισεκατομμυρίων για την ενέργεια. Κάτι που αντιστοιχεί σε διπλασιασμό της ισχύω του τρέχοντος μηχανισμού συνδέοντα την Ευρώπη. Αλλά σας διαβεβαιώ ότι αυτή η βελτίωση ήταν απολύτω απαραίτητη. Και φυσικά είναι ώρα τώρα να ε, επαναθεωρήσουμε και τις προτεραιότητές μας και να τις επικαιροποιήσουμε. Είπα στην αρχή της παρουσίασής μου πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση με το φυσικό αέριο και πόσο σημαντικό είναι να εξασφαλίσουμε ένα επαρκές επίπεδο διαφοροποίησης. Διαφοροποίησης και των προμηθευτών αλλά και των διαδρόμων. Επίσης θα πρέπει να ε, δράσουμε τους, τα κενά που έχουμε, να διορθώσουμε τα κενά που έχουμε και στις υποδομές αλλά και στην καινοτομία. Θα πρέπει να διορθούν αυτά τα κενά, αλλά οι νέες μας προτεραιότητες μας αφορούν ε, σχέδια ηλεκτρισμού, ηλεκτροδότησης, αλλά και το νέο παράθυρο για να καλύψουμε και σχέδια ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που έχουν διασυνοριακή σημασία. Το τέστην τώρα μπορούμε να επικεντρωθούμε περισσότερο στις μελλοντικές δαπάνες και στο τι μελγενέστε. Σίγουρα οι μελλοντικέ δαπάνε θα πρέπει να διορθώσουν τα υπάρχοντα κενά στι διασυνδέσει. Γιατί έχουμε ακόμη 10 κράτη-μέλη που είναι κάτω του 10% της ε, διασύνδεσης στην Ευρώπη. Επίσης, είναι εξίσου σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι αυτή τη στιγμή είμαστε η μόνη ε, μεγάλη οικονομία του κόσμου που ε, το 30% της ηλεκτρικής ενέργειας το παράγει από ΑΠΕ, από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και την επόμενη δεκαετία αυτό το 30% θα γίνει πάνω από 50%. Κατά συνέπεια θα αυξηθεί η ανάγκη εισαγωγής και εξαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας γιατί η κατάσταση ε, μεταβάλλεται ανάλογα με τις καιρικέ συνθήκες και τις ε, ικανότητες παραγωγής, ε, γιατί έχουμε υδροελεκτρική ενέργεια, αιωλική ενέργεια και μάλιστα αιωλική onshore και offshore. Και η ανάλυση μας είναι ξεκάθαρη. Δεν θα εμείνουμε στο πλαίσιο ε, της ανταλλαγής ηλεκτρονικής ενέργειας, ε, ηλεκτρικής ενέργειας μόνο. Και στο πλαίσιο αυτό θα έχει κέρια σημασία να θέσουμε τέρμα σε κάποιες απαράδεκτες καταστάσεις. Και αυτό θα πρέπει να το φροντίσουμε με τις ενέργειές μας. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε ακόμη τρεις χώρες κράτη, τρεις ε, χώρες μέλη που ε, εξακολουθούν να εξαρτώνται από το ρωσικό δίκτυο. Και βρισκόμαστε στο 2018. Αυτές οι χώρες έχουν ε, προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2004 και συνεργαζόμαστε όλοι μερείς και όλο νύχτη για να βρούμε μαζί με την Πολωνία για παράδειγμα τρόπο να συγχρονίσουμε την Πολωνία και τις ε, βαλτικές χώρες ώστε να μειωθεί η εξάρτησή τους από το ρωσικό δίκτυο. Γνωρίζετε όμως την ιδιάζουσα κατάσταση που έχουμε με την ενεργειακή νησίδα που αποτελεί η Βυρική Χερσόνησος. αυτή η ενεργειακή απομόνωση της Ιβερικής Χερσονήσου μας απασχολεί. Με το νέο σχέδιο όμως που έχουμε θα καταλήξουμε σε ένα επίπεδο άνω το 80% διασύνδεση μεταξύ Ισπανίας και Γαλλίας. Αυτό θα είναι θεμελιώδες βήμα πρόοδου για να τεθεί ένα τέρμα σε αυτή την ενεργειακή απομόνωση της Ιβηρικής Χερσονήσου. Και προσπαθούμε να οργανώσουμε μια νέα σύνοδο κορυφής, το συντομότερο δυνατό, μεταξύ ε, Γαλλίας, Ισπανίας, Πορτογαλίας και Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα θέματα αυτά, για να τεθεί ένα τέρμα στην ενεργειακή απομόνωση της Ιβηρικής Χερσονήσου. Πάντως, εξακολουθούμε να επιμένουμε στην αύξηση του επίπεδου διασύνδεσης, όχι μόνο στο 10%, όχι μόνο κατά 10% μέχρι το 2020, Μέχρι το 2020 όλα τα κρατη και πιστεύω ότι όλα τα κρατη θα έχουν φτάσει σε αυτό το 10%, αλλά θέλουμε να ξεπεράσουμε αυτό το 10%, να φτάσουμε σε 15% διασύνδεσης, κάτι που θα αποτελέσει ένα ουσιώδες νέο βήμα πρόοδο. Αλλά όπως είπα θα προτείνουμε και μέτρα για να ανταποκριθούμε στα αιτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στο ψήφισμά σας στις 13 η Μαρτίου του 2018. Γι' αυτό προτείνουμε επέκταση του μηχανισμού συνδέοντας στην Ευρώπη, του νέου ΣΕΦ, για να καλύψει και τις διασυνοριακές ε, εξελίξεις. Και με την νέα οδηγία για τα ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έχουμε στόχο με την υποστήριξη του ε, εισηγητή σας να δημιουργήσουμε μια ευρύτερη αγορά που θα ξεπερνάει τα εθνικά σύνορα γιατί το κόστος μειώνεται και η μείωση του κόστους για τις ΑΠΕ είναι εντυπωσιακή. Ιδιαίτερα την τελευταία διότι έχει μειωθεί αισθητά το κόστος των ΑΠΕ και όταν πριν από δυόμιση χρόνια εγκαινιάσαμε την πρωτοβουλία για τη Βόρεια Θάλασσα, το κόστος ήταν 150 ευρώ ανά μεγαβάτ για τις μεγάλες ε, ανεμογεννήτρες offshore μετά, δύο, δύο χρόνια μετά και λίγους μήνες, δύο χρόνια και λίγους μήνες μετά τη τελευταία καταμέτρηση, το κόστος έχει πέσει περίπου στο, στα 60 ευρώ ανά μεγαβάτ, από 150. Μερικές φορές το ζητούμε την ενέργεια, σκεφτόμαστε μόνο το μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Αλλά τώρα είμαστε σε μια κατάσταση όπου η καινοτομία και η νέα βιομηχανική βάση καθαρής ενέργειας, ιδιαίτερα για τις μεγάλες ανεμογεννήτριες, δείχνουν τι δυνατότητα υπάρχει για την, για την ανάπτυξη μιας πραγματικά ανταγωνιστικής προσέγγισης για τις ΑΠΕ. Και αυτό ισχύει και για την ελληνική ηλιακή ενέργεια, αλλά όλο και περισσότερο για την αιωλική ενέργεια, ακόμη και για την offshore αιωλική ενέργεια. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι θα διασφαλίσει την τεχνολογική ηγετική της θέση με όλες τις εγκαταστάσεις αυτές που έχει σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό είναι θεμελιώδες και θα το προωθήσουμε. Επίσης, θα αναπτύξουμε όλες τις μεθοδολογίες που χρειαζόμαστε για να εφαρμόσουμε αυτές τις προσπάθειες τους επόμενους μήνες, γιατί διαβλέπουμε μεγάλο δυναμικό αύξησης της συνολικής μας ικανότητας, προκειμένου να αξιοποιήσουμε αυτό το νέο παράθυρο ευκαιρίας. Χάρη σε ένα αυξημένο επίπεδο και περιφερειακής συνεργασίας. Γνωρίζουμε όλοι ότι ο μηχανισμός περιφερειακής ικανότητας είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Πηγαίνουμε παντού στην Ευρώπη. Αναφέρθηκα στην κατάσταση που έχουμε μεταξύ Πορτογαλίας και Ισπανίας, αλλά μπορώ να σας αναφέρω και άλλο παράδειγμα την Κεντρική Ευρώπη και την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Δεν είναι τόσο γνωστό το παράδειγμα, αλλά πολλές από τις χώρες αυτές έχουν φτάσει ε, και έχουν υλοποιήσει τους στόχους τους για τις ΑΠΕ ε, για το 2020. Και το έχουμε αυτό στο Δούναβι, στην Πολωνία, στη Βαλτική. Είχαμε επευκαιρία πολύ σημαντική συζήτηση και μάλιστα τον περασμένο μήνα είχαμε και μια εκδήλωση στο Κατοβίτσε και το κάναμε και στην Νοτιοανατολική Ευρώπη αυτό. Και ελπίζω με τη νέα πρόταση να είμαστε καλά εξοπλισμένοι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να προλάβουμε και τις εξελίξεις εν ώψη του επόμενου ΠΔΠ και θα με κρατήσουμε την επαφή μας για να είμαστε πάντα ενήμεροι για τις νέες προτεραιότητες. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για την παρουσίασή σας και τώρα πρώτος να μιλήσει ο εισηγητής μας, η εισηγητρία μάλλον για το συνδυόντα στην Ευρώπη, κυρία Βυρκούνεν. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εσάς κύριε Γενικέ Αριστόρη για τα όσα μας είπατε. Είναι πολύ σημαντικό πρόγραμμα αυτό για την Ευρώπη και για την Επιτροπή μας γιατί ε, ένας από τους στόχους μας είναι να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη, στην ανταγωνιστικότητα, στην απασχόληση και το συνδύοντα στην Ευρώπη να ρίξει κανεί τη μεσοπρόθεσμη αξιολόγηση του προγράμματο. Ε, καταλήξαμε στο ότι είναι πολύ πετυχημένο αυτό το πρόγραμμα, οπότε τώρα εξετάζουμε την ψηφιοποίηση, την ενεργειακή πολιτική, είμαστε συναρμόδιοι με την ε, τρανς και την ε, και η δική μας επιτροπή τέλος πάντων. Ε, οπότε η δουλειά μας θα παρουσιάζει ενδιαφέρον στο μέλλον. Οπότε το Κοινοβούλιο με την Επιτροπή μας έχει εξετάσει το θέμα της Ενεργειακής Ένωσης να δούμε πώς θα έχουμε βιωσιμότητα, πώς θα έχουμε αποτελεσματικότητα στην ενεργειακή αγορά της Ευρώπης, οπότε χρειαζόμαστε αυτά τα αξιόλογα εργαλεία μέσα πολιτικής γιατί ε, έχουμε αυτές τις προτεραιότητες που μας παρουσιάσατε κύριε Γενικέ, τα οποία είναι στο ίδιο μήκο κύματο με τις δικές μας ε, συζητήσεις. Εκεί επιστρέφουν το ενδιαφέρον μας, δεν θα πρέπει επομένω να υπάρχουν κενά στην πολιτική μας αυτή, εάν θέλουμε να υπάρξει και στην ενεργεια ενιαία αγορά. Οπότε θα πρέπει τώρα να προσέξουμε τις ενέργειες τις διατομιακές, γιατί μία από τις κεντρικές ιδέες του θέματος είναι ότι όταν κανείς τα συνδυάζει μεταφορές, ενέργεια, ψηφιοποίηση, τότε προκύπτουν οι συνέργειες όπως τα εφή δίκτυα, η υποδομή για τα καύσιμα, ε, για τις μεταφορές, για αυτοματοποιημένη, αυτόματη τέλος πάντων κινητικότητα και κυβερνοασφάλεια. Οπότε έχουμε όλους αυτούς τους ε, τομείς και με την ψηφίπηση και με την κινητικότητα θα πρέπει να εξετάσουμε το πώς θα έχουμε τέτοιες συνέργειες διατομιακές και νομίζω ότι η Επιτροπή μας συμφωνεί με αυτές τις προτεραιότητες της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής για όλα αυτά τα θέματα. Οπότε, όπως έχουμε εντατική δουλειά μπροστά μας σε επόμενες εβδομάδες, γιατί θα πρέπει να ετοιμάσουμε με τους ε, συνεισηγητές αυτή την ε, έκθεση σε τρεις-τέσσερις εβδομάδες ε, μαζί με την Επιτροπή Μεταφορών. Είναι δική μας προτεραιότητα επίσης. Θέλουμε να τα πάμε καλά. Θέλουμε να τα πάμε καλά και στις διαπραγματεύσεις. Να ξεκινήσουμε με το δεξί. Το φθινόπωρο Και βέβαια περιμένω πως και πως να ακούσω τι έχουν να πούν οι συνάδελφοι και οι σίγουρος που θα είναι ενδιαφέρουσες στις συζητήσεις μας. Όλοι οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση αυτή έχουν υψηλές προσδοκίες, γιατί υπάρχουν κενά στην πολιτική μας. Και να έχουμε για την ενεργή ασφάλεια επενδύσεις και για να είναι αποτελεσματική η αγορά ενέργειας θα πρέπει επίσης κάτι να κάνουμε για τα δίκτυα σε όλη την Ευρώπη. Ευχαριστούμε κυρία Λέω Πρόεδρο. και τώρα. Οι σκιώδες εισηγητέ έχουν τον λόγο. Για το συνδύο. κυρία Κουμπούλα Νάτρη. Ευχαριστώ. Νομίζω έχει, ότι έχει μέλλον αυτή η πρόταση. Ενθαρρυντικά τόσο μα είπε η Κομισιόν και την ευχαριστούμε. Ε, επίσης, και τα ψηφιακά είναι αρμοδιότητά μας, όπως είπε η συγκήτρια, οπότε έχουμε όλα αυτά τα ωραία θέματα να εξετάσουμε από κοινού με την Επιτροπή Μεταφορών και τις μεταφορές βέβαια, άρα έχει μέλλον υπόθεση. Και γνωρίζουμε ότι και το αυτό θα είναι πάρα πολύ σημαντικό, το κλίμα, η υπόθεση για το κλίμα μετά το Παρίσι και η Ευρώπη θα πρέπει να τα καταφέρει σε αυτό το μέτωπο. Θα πρέπει επίσης να επιταχύνουμε τις ενεργειές μας όσον αφορά την κλιματική αλλαγή. Και θα πρέπει επίσης να τα λάβουμε αυτά υπόψη μας. Εγώ θα ήθελα να μπω στις λεπτομέρειες ε, δηλαδή το πώς ακριβώς ε, πρέπει να εξετάσουμε αυτό το 65% που δαπανάτε, αν θα πρέπει να δαπανάτε για θέματα κλίματος. Ε, θα ήθελα να ακούσω τους συναδέλφους να μας πούν και αυτοί πώς ορίζουν το όλο θέμα. Και νομίζω ότι τώρα πλέον ε, πρέπει να δοθούν κονδύλια και για τις ε, διασυνοριακές απέ. Ναι, είναι τοπικό το θέμα, αλλά πρέπει να εξετάσουμε και το θέμα των ε, δικτύων. Πρέπει να το εξετάσουμε και αυτό. Όσον αφορά τώρα στην ηλεκτρική ενέργεια ως προτεραιότητα, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αν δούμε τα οχήματα, αν δούμε τους υπολογισμούς, το πόσο μπορεί να υπάρξει βελτίωση, εξαρτάται βέβαια και το πώς προσφέρονται άλλες μορφές ενέργειας. Ε, οι εκπομπές. Κάπου είναι 30%, κάπου 70%. Εξαρτάται λοιπόν και από το πώς μπορούμε να αντικαταστήσουμε την ηλεκτρική ενέργεια με άλλες μορφές ενέργειας. Αυτή τη στιγμή ε, νομίζω ότι ε, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε το θέμα της ε, θέρμανσης, γιατί αν συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε ως θερμαντικά στοιχεία ιδιαίτερα ρηπογόνα, τότε νομίζω ότι η Ευρώπη δεν θα τα καταφέρει καλά. Εγώ θέλω να ελπίζω ότι θα περάσει το πρώτο πακέτο για την καθαρή ενέργεια ε, το Κοινοβούλιο να συνεχίσει με το Συμβούλιο να εργάζεται προς αυτήν την κατεύθυνση και κυρίως όσον αφορά τις ε, περιφερειακές αγορές ε, ενέργειας. Εμείς οι Βόροι ξέρουμε ότι λειτουργεί το θέμα. Πολλές χώρες Βαλτικής πάνε μαζί μας, η Εστονή, παραδείγματο χάρη. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα. Προσβλέπω λοιπόν στη μελλοντική συνεργασία. Σας ευχαριστώ από τους συντηρητικούς μεταρρυθμιστές το λόγο ο κύριος Τσέσακ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον Γενικό Διευθυντή για την ανάλυση που μας έκανε στην παρουσίασή του. Θα ήθελα πρώτα να συγχαρώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί ε, φρόντισε να παραμείνει στον προηγούμενο προϋπολογισμό, να μην τον περικόψει. Ε, γνωρίζουμε ότι το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο είναι η βάση ε, για τα θέματα αυτά και σίγουρα ε, το συνδέοντα στην Ευρώπη θα είναι από τους πιο αποτελεσματικούς μηχανισμούς. Θα πρέπει λοιπόν να διαφυλάξουμε αυτό το νευραλγικό πρόγραμμα για την εξασφάλιση σημαντικών υποδομών και για την ενεργειακή ασφάλεια. Ε, το Συνδέοντα στην Ευρώπη ε, χρηματοδοτεί πολλά σχέδια, όπως τον, φυσικό, τον αγώ φυσικού αερίου στη Βαλτική, όταν εξετάζουμε το Nord Stream 2 ή την απεξάρτηση από, τη, από το ρωσικό φυσικό αέριο. Γι' αυτό χρειαζόμαστε τέτοια προγράμματα και επαρκή χρηματοδότηση. Έχω κάποιες ερωτήσεις. Στις Βρυξέλλες ε, συζητούμε το θέμα της ηλεκτροκίνησης και ε, οι συζητήσεις πάντα καταλήγουν στα ίδια συμπεράσματα στα ίδια ερωτήματα. Θα πρέπει να αναπτύξουμε υποδομές ε, για την ε, εξυπηρέτηση αυτών των αυτοκινήτων ή να επικεντρωθούμε περισσότερο στην παραγωγή περισσότερων ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Θα πρέπει πρώτα να λύσουμε το ζήτημα των σημείων επαναφόρτηση των ηλεκτρονικών οχημάτων. Θα πρέπει να διευκολύσουμε και τη διάθεσή του στην αγορά το συντομότερο δυνατόν. Δεν θα πρέπει να χάσουμε αυτή τη σημαντική ευκαιρία. Με βάση του τελευταίου υπολογισμού τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, λίγε προσπάθειε έκαναν τα κράτη-μέλη για την αύξηση των ηλεκτρικών οχημάτων. Το αναφέρατε κι εσεί ε, ε, κύριε Γενική Διευθυντά. Ένα από τα σημαντικότερα προσκόμματα είναι το κόστος των σημείων επαναφόρτησης. Το συνδέοντα στην Ευρώπη μπορεί να προσελκύσει δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις προκειμένου να δημιουργηθούν περισσότερα σημεία επαναφόρτηση. Επίσης, το ζήτημα της συνέργειας. Θα μπορούσατε να μας πείτε τι έγινε προκειμένου να βελτιωθεί η διατομιακή συνεργασία ε, στα θέματα αυτά. Γιατί είναι σημαντικό να αξιοποιήσουμε την τεχνογνωσία και να αναπτύξουμε ε, έξυπνα δίκτυα, δίκτυα. Είναι πολύ σημαντικό και κυρίως ε, να δούμε πώς αυξήσουμε την ηλεκτροκίνηση. Επίσης, να μην ξεχάσουμε την ψηφιακή λειτουργία των σημείων επαναφόρτησης. Ε, πώς μπορούμε να συνδυάσουμε τον συνδέοντα στην Ευρώπη με άλλα, με άλλα προγράμματα όπως το Ορίζοντας Ευρώπη. Επίσης, πώς θα βελτιώσουμε τη διασύνδεση μεταξύ Πολωνίας και Βαλτικών χωρών με την υπόλοιπη Ευρώπη. Πώς το συνδέοντας την Ευρώπη θα διευκολύνει την διασυνοριακή διασυνδεσιμότητα. Επίσης, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν σκοπεύετε να ενισχύσετε τα εθνικά δίκτυα φυσικών αερίων ώστε να μειωθεί η επιβάρηση ή να αυξηθεί ε, το ποσοστό των ΑΠΕ. Γιατί πολύ συχνά μιλούμε ότι δεν έχουμε interconnectors ε, αρκετούς, αλλά μερικές φορές αυτό το θέμα το συνδέουμε με μόνο μια χώρα, χωρίς να λαμβάνουμε μια πιο σφαιρική προσέγγιση. Σας ευχαριστώ. Πολύ σημαντικά τα ερωτήματα που θέσατε, κύριε συνάδελφε. Ο κύριος Πέτερσεν έχει τώρα το λόγο και μέρος των φιλελευθέρων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, Ντομινίκα, για τις ε, παρατηρήσεις σας. Ε, πρέπει να σας πω ότι μας αρέσει πάρα πολύ που αποδείτε ιδιαίτερη σημασία στο τι θα γίνει με τη Συμφωνία των Παρισίων από 5,3 σε 8,7 δις αυξήθηκε ε, το όλο χαρτοφυλάκιο του συνδέοντος στην Ευρώπη. Αποδείχθηκε ότι πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό πλαίσιο ε, για να ε, αυξηθούν και οι ιδιωτικέ και οι κρατικέ επενδύσει. Και βλέπουμε ότι το 60% του νέου προπολογισμού για το συνδέοντα στην Ευρώπη ε, προβλέπεται στο να περιοριστούν οι εκπομπέ αερίων. Σα λέω, χρειάζονται φιλόδοξοι στόχοι σε αυτό τον τομέα. Και εμεί συμφωνούμε ότι πρέπει να βελτιωθεί η διασυνοριακή υποδομή, να προβληθούν περισσότερο οι ΑΕΠ σε αυτό το ενεργειακό μείγμα, κυρίω όσον αφορά το στόχο στόχο του να ανέλθουν στο 22% μέχρι το 2030. Επιτρέψτε μου να κάνω κάποιες ε, κρίσιμες ε, μορφής ε, παρατηρήσεις. Δηλαδή, αν τελικά πρόκειται να επιτύχουμε μια κοινωνία χωρίς εκπομπές άνθρακα μέχρι το 2050, αν το θέλουμε αυτό πρέπει να αποδώσουμε προτεραιότητα στις υποδομές ε, για την ενέργεια. Και η έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης ε, του Ιουλίου του 2017, εκεί αναφέρεται ότι το 65% των επενδύσεων για τη μετάβαση προβλέπονται ακριβώς ε, στον τομέα της ενέργειας. Και αυτό εφόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί να επιτύχει το στόχο της. Στα άρθρα 7, 90 και 30 αναγράφονται τα κριτήρια και εξ όσων γνωρίζω αναφέρεται ότι μέχρι το Δεκέμβρη του 2019 η Κομισιόν πρέπει να εγκρίνει μια κατεξουδότηση πράξη που θα ε, αναφέρει τα επόμενα κριτήρια που πρέπει να στηριχτούν. Εγώ προτείνω η Κομισιόν να αναθεωρήσει τα κριτήρια που υπάρχουν τώρα, που αναφέρονται στο άρθρο 14 και στο παράρτημα 2 του τρέχοντος κανονισμού για το συνδέοντα στην Ευρώπη. Αυτά τα κριτήρια ε, θα επιτρέψουν ε, μάλλον τώρα τα κριτήρια επιτρέπουν να γίνονται πολλές επενδύσεις στα ορυκτά καύσιμα και εγώ πιστεύω ότι στα νέα κριτήρια πρέπει να επισημαίνεται ότι πρέπει να μειωθούν οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και να εφαρμοστεί η συνθήκη των Παρισίων και να ληφθεί υπόψη και το μειωμένο κόστος των ΑΕΠ από το 30 και μετά. Και μόνο έτσι ο μηχανισμός ε, συνδέοντας ε, την Ευρώπη πραγματικά θα συμβάλλει στην Ενεργειακή Ένωση. Θέλω πολύ να ακούσω τις παρατηρήσεις σας, ε, κύριε Ριστόρη, σχετικά με αυτά τα κριτήρια για το πώς μπορούμε να επιτύχουμε όλους αυτούς τους στόχους τους οποίους επιδιώκουμε. Πολύ ωραία. Επόμενος ε, εκ μέρους των Πρασίνων, ο κύριος Μαρτσέλεση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και το Γενικό Διευθυντή Ριστόρη για τις εξηγήσεις που μας έδωσε και την παρουσίαση που έκανε. Ε, πολλά θετικά ως προς τα διασυνοριακά προγράμματα, για παράδειγμα, ή τις συνέργειες που μπορούν να δημιουργηθούν μεταξύ διαφόρων τομέων ή καλύτερο συντονισμό που προβλέπεται μεταξύ ε, των διαφορετικών ταμείων, των επενδυτικών ταμείων, των ορίζοντα με το συνδέοντα στην Ευρώπη. Τώρα, έχω κάποιες επικρίσεις ως προς την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά τα θετικά φαίνεται ότι υπάρχει μια αιμονή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, στα σχέδια φυσικού αερίου ε, που μονοπολεί περισσότερο συνήθως τα σχέδια κοινού ενδιαφέροντος ε, επίσης, τι γίνεται με τις υποδομές, ε, με ε, τους αγωγούς διοξιδίου του άνθρακα, όπως θα λέγαμε. Για αυτά τα θέματα έχουμε κάποιες επιφυλάξεις. Επίσης, ό,τι αφορά τη διασύνδεση που προτείνει, στη Βισκάγια, για παράδειγμα, και εκεί έχουμε πολλές αμφιβολίες για το κατά πόσο είναι ε, σκόπιμος ένας τέτοιος αγωγός και ποιο θα είναι το οικονομικό κόστος για την Ισπανία, η οικονομική επιβάρηση της Ισπανίας ή το επίπεδο συμμετοχής ή διαφάνεια που μπορεί να εξασφαλιστεί γιατί έχουμε στο Βασκονικό κόλπο δύο πλευρές ε, και στην Ακητέν και στη, στη χώρα των Βάσκων, οπότε εκεί ε, θα πρέπει να ταχθούμε υπέρ της διασύνδεσης, αλλά όχι πάση θυσία ούτε με ε, κάθε τρόπο και χωρίς διαφάνεια. Έχω κάποιες ερωτήσεις για τις προτάσεις σας. Η πρώτη αφορά τη τον κανονισμό για τα διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας. Ε, ο κανονισμός έγινε το 2013. Στο μεταξύ είχαμε τη Συμφωνία των Παρισίων. Δεν ξέρουμε πώς αναθεωρήθηκε ο κανονισμός, ε, έχει επικαιροποιηθεί προκειμένου να συμβαδίζει με τη Συμφωνία των Παρισίων που αλλάζει τελείως τα δεδομένα. Επίσης, πότε σκοπεύετε να αναθεωρήσετε αυτό τον κανονισμό που ανάγεται στο 2013 για τα ΤΕΝ ή για τα διευρωπαϊκά δίκτυα Σε Ό,τι αφορά την ανανέωση του ΣΕΦ, είπατε ότι τα περισσότερα σχέδια του συνδέοντα στην Ευρώπη θα πρέπει να αφορούν ε, τους ε, διαδρόμους ηλεκτρικής ενέργειας είπαμε ε, μέχρι 90% ε, των ε, κονδυλίων θα πρέπει να πηγαίνει σε θέματα ηλεκτρικών δικτύων, αλλά τίποτα συγκεκριμένο δεν προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι ακριβώς επίπεδο είναι το ζητούμενο, θα πρέπει να το ποσοτικοποιήσετε. Αυτά και τέλος για το mainstreaming. Αναφερθήκατε στο 60%. Δεν αρκεί όμως αυτό, γιατί το 24 είναι σημαντικό, το COP24 είναι σημαντικό, γιατί θα είναι η συνέχεια της Συμφωνίας των Παρισίων. Επίσης, στην επόμενη ε, έκθεση για το EPCC θα δούμε ότι δεν πάμε καλά σε ό,τι αφορά το στόχο της μη υπέρβασης αύξησης θερμοκρασίας κατά κανένα μισή βαθμό. Θα πρέπει να έχουμε 100% συνεκτίμηση της διάστασης του κλίματος, το climate mainstreaming. Αν θέλουμε να είμαστε παγκόσμιοι ηγέτες στην καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών, θα πρέπει το climate mainstreaming, τη συνεκτίμηση του κλίματος στις πολιτικές μας, να το έχουμε πλήρως Αυτά. Ευχαριστώ. Τώρα περνάμε στους υπόλοιπους α, ομιλητές. Η κυρία Βέρνερ, ευχαριστώ πολύ πρόεδρε και ευχαριστώ και Ριστόρ για την ε, πολύ καλή σας έκθεση. Εννέα δις για το συνδέοντο στην Ευρώπη είναι μια πολύ καλή είδηση. Και εγώ αναφέρομαι στην ενέργεια, πιο συγκεκριμένα στην ηλεκτρική ενέργεια. Είπατε Είπατε κράτη-μέλη και ε, πολλά από αυτά στη διασύνδεση είναι κάτω από 10%. Προφανώς και πρέπει να αυξηθεί το ποσοστό. Αν θα αρκεί το 15% αυτό δεν το ξέρουμε. Ίσως και αυτό το 15% να είναι λίγο. Γιατί ε, αν δούμε την ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας χρειαζόμαστε μη μεγάλη ε, αγορά με ρευστότητα. Πρέπει να έχουμε κατά νου και το εμπόριο. Και το εμπόριο λειτουργεί σε διασυνοριακή βάση. Γι' αυτό λοιπόν η διασύνδεση είναι η μισή αλήθεια. Να δούμε και πίσω από αυτό, να δούμε τι κρύβεται πίσω από τη διασύνδεση. Δηλαδή, τα κράτη-μέλη είναι σε θέση να παίρνουν ε, ρεύμα από άλλες χώρες και να το διανέμουν στη δική τους την επικράτεια. Γιατί εκεί μιλάμε για αποκεντρωμένα δίκτυα διανομής που πρέπει να βελτιωθούν. Νομίζω ότι εκεί η πολιτική λυπόμεθαν κατά πολύ, γιατί το θέμα δεν είναι μόνο να φτιάξει κανείς το μηχανισμό και το δίκτυο που είναι πίσω από τα σημεία σύνδεσης θα πρέπει να είναι συμβατό. Νομίζω λοιπόν ότι σε ορισμένα κράτη-μέλη λείπει η προθυμία να βελτιωθούν τα δίκτυα. Τίθεται λοιπόν το ερώτημα τι ακριβώς μπορεί να κάνει η Επιτροπή, γιατί αλλιώ ξέρετε κάτι, θα έχουμε ένα τεράστιο δυναμικό στα σημεία διασύνδεσης, αλλά δεν θα μπορούμε να το διανύμουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η κυρία Γκροστέτ έχει το λόγο. Να ευχαριστήσω τον Ντομινίκ Ριστορή. Είναι σπουδαία η δουλειά που κάνει, ιδιαίτερος χρήσιμη για μας. Να πούμε για τις διασυνδέσεις στα κράτη-μέλη, οπότε έτσι κυκλοφορεί καλύτερα η ενέργεια και για να μπορέσουν να είναι βιώσιμες θα πρέπει να εξασφαλιστεί το να είναι επικερδές, βράχη και μακροπρόθεσμα. Και έτσι θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τα έργα, τα προγράμματα αυτά, πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις, δεν ξέρω αν κάνω λάθος, αλλά μου φαίνεται ότι αυτό δεν λαμβάνεται τόσο πολύ υπόψη. Πέστε μας, σας παρακαλώ, κάνετε αυτή την ανάλυση κόστους-οφέλους για την επιλογή των έργων και προγραμμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μπορείτε να αναβαθμίσετε αυτή την ανάλυση και μετά να θεωρήσετε κοινό ενδιαφέροντος κάποιο έργο πρόγραμμα και να μπορούμε στο μέλλον να κάνουμε τη σχετική πρικοδότηση. Ευχαριστούμε πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Μπλάνκο Λόπεθ, συναδελφοί, έχει λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Το πρόγραμμα στην Ευρώπη είναι πολύ σπουδαίο και έχει σχέση με την ενέργεια. Άρα το σούτο μάλλον απαραίτητο, γιατί θέλουμε να φτιάξουμε μια ενεργειακή ένωση και έτσι να υπάρξει περισσότερη αυτονομία στην Ευρώπη, λιγότερη εξάρτηση. Αυτός είναι ο, ρόλος, ο στόχος των διασυνδέσεων. Αυτό θέλουμε. αυτό είχαμε κατά νου όταν προσπαθούσαμε και ευχαριστούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη δουλειά της, για τις συμφωνίες αυτές που έκλεισε και να υπάρχει αυτή η φιλόδοξη οδηγία για τις ανέργειε πηγές ενέργειας, ούτω ώστε να μπορέσουμε να προωθήσουμε τις καθαρές ενέργειες και αυτό θα, θα είναι η ατμομηχανή για να φτάσουμε στην αυτάρκεια στην Ευρώπη. Οπότε γι' αυτό και είχαμε αυτή την ε, τροποποίηση, την τροπολογία τέλο πάντων για να έχουμε τέτοιες διασυνδέσεις, για να φτάσουμε σε τέτοιο πλαίσιο πολιτικής καθαρών ενεργειών στην Ευρώπη. Μπράβο για αυτή την πρωτοβουλία. Έτσι φτάνουμε πιο κοντά στο στόχο που έχουμε για περισσότερη ενεργειακή ε, αυτάργεια και για πρόθεση των, ε, της που για το μέλλον που είναι η καθαρή ενέργεια. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κύριε Ριστορή. Και, λέει κύριος Μαρτίν, είναι προτεραιότητα το, για τις διασυνδέσεις, ιδίως όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια, κάτι πολύ θετικό. Όπως γνωρίζετε, υπάρχει πρόβλημα. Ιστερούμε όσον αφορά τον ε, στόχο ε, της COP21. Τα είπε και ο συνάδελφος Μαρσελέση, γιατί θα πρέπει να μην επικεντρώμαστε μόνο στο φυσικό αέριο, γιατί έτσι λέει η ρυθμιστική αρχή στη Γαλλία, ότι ο αγωγός του Ροδανού ε, συνδέει Ισπανία, Γαλλία, αλλά ήδη το, το θέμα έχει ε, πάρει υπερβολικές διαστάσεις. Ε, πολλές δαπάνες. Μα όμως ε, σε τέτοιες εποχές αυτό δεν είναι τόσο καλό. Θα μας κατηγορήσουν ε, την επαύριο οι Ευρωπαίοι για διασπάθηση του χρήματος, γιατί υπάρχουν άλλες προτεραιότητες. Τι γίνεται με το κλίμα. Ακόμα κάποια κρατή υστερούν πάρα πολύ όσον αφορά την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας. Ξέρω ότι είναι κυρίως μου αλλά θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με κάποιες περιοχές που είναι πιο φιλόδοξες, ε, πιο εφάνταστες από ότι οι κεντρικές κυβερνήσεις και ε, αν υπάρξει χρηματοδότηση μπορούμε να προχωρήσουμε σε, στην ενέργεια που θέλουμε. Ο κύριος Τούρμες, ευχαριστώ Ντομινίκ και ευχαριστώ τη, το, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Επιτελείο της γενική Γενικής Διεύθυνσης για την πολύ καλή πρόταση ε, το Συμβούλιο θα προσπαθήσει να περικόψει το μισό τη προτάσεις σα ε, Για να το αποφύγουμε θα πρέπει να κάνουμε δύο να Ευχαριστώ καταρχήν την κυρία Βίρκουνεν, την εισηγήτρια, που αναφέρθηκε στο γεγονό ότι θα πρέπει να δώσουμε μια βιομηχανική διάσταση στην πρόταση. Η Ευρώπη με, η Ευρώπη με τη Siemens, ε, με την ABB, με τις νεοφυείς, ε, νεοσύστητες επιχειρήσεις που έχουμε για, τους, για τα σημεία επαναφόρτησης, θα μας βοηθήσουν να δημιουργήσουμε μια αγορά του μέλλοντος ε, το ψηφιακό συναντά τις μεταφορές και την ενέργεια. Θα πρέπει να τονίσουμε αυτή την αλληλεπίδραση. Και για να καταρρύψουμε το επιχείρημα του Συμβουλίου που θα θέλει να μειώσει τον προϋπολογισμό, θα πρέπει να έχουμε διάστητα επιχειρήματα. Οι βαλτικές χώρες έχουν για γεωπολιτικούς λόγους ε, να, να απεξαρτηθούν από τη Μόσχα και να συγχρονιστούν με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ισπανία και η Πορτογαλία θα γίνουν από τι μεγαλύτερε εξαγωγέ ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ στο μέλλον. Οπότε συμφωνώ ότι θα, ε, θα έχουμε ένα καλώδιο μεταξύ Λιθουανίας και Πολωνίας και χάρη σε αυτό θα μπορούμε να έχουμε ολική ενέργεια στην θάλασσα. Επίσης, ε, ε, και στην Εστονία, Λιθουανία, Εστονία έχουμε σημαντικά σχέδια για αιωλική ενέργεια offshore. Θα μπορούσαμε λοιπόν να έχουμε μια πραγματικά διασύνδεση στις χώρες αυτές. Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η Ρουμανία είναι πιθανώς εξαγωγές αιωλικής ενέργειας ε, και πήγες και με θαλάσσιες ανεμογεννήτριες. Επίσης στην ε, Βόρεια Θάλασσα έχουμε σημαντικό κοίτασμα και από τη στιγμή που θα υπογραφεί το διαζύγιο με, το, με την Μεγάλη Βρετανία, θα έχουμε το σχέδιο Don't Go Back. Στην Βόρεια Θάλασσα, μεταξύ πέντε χωρών, έχουμε μια περιοχή που δεν έχουμε ούτε 30 μέτρα βάθος. Εκεί θα μπορούσαμε κάλλιστα να δημιουργήσουμε αιωλική ενέργεια 500 και μεγαβάτ και θα μπορούσαμε ε, να παράγουμε πράσινο υδρογόνο στην υπηρετική Ευρώπη. Θα έχουμε λοιπόν πολλά ενδιαφέροντα για τις κυβερνήσεις ε, προγράμματα και σχέδια και έτσι μπορούμε να δημιουργήσουμε μια πλειοψηφία στο Συμβούλιο ώστε να διαφυλάξουμε τον προϋπολογισμό προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ κυρία Πιλάρ Δελκαστίγιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον Ντομινί Κριστορή, τον Γενικό Διευθυντή που ήρθε για να μας κάνει την παρουσίαση. Εγώ θα σταθώ ε, μόνο όπως έκανα καθόλου τη διάρκεια της συζήτησης και της υποβολής των τροπολογιών στο θέμα της διασύνδεσης για την ηλεκτρική ενέργεια. Μας είπε η κυρία Γκροστέτ ότι θα πρέπει να δούμε το λόγο κόστους οφέλους. Φυσικά να δούμε το, τη σχέση κόστους οφέλους, αλλά με μία μακροπρόθεσμη ε, προσωμείωση και προοπτική, όχι μόνο ε, υπό το πρίσμα της βραχυπρόθεσμης ή της άμεσης ε, ε, αξιοποίησης και άμεσου κέρδους. Και από αυτή την άποψη είναι σημαντικό να συνδέσουμε την ανάπτυξη των υποδομών με την υλοποίηση των στόχων. Όσο μεγαλύτερη φιλοδοξία έχουμε σε θέματα ΠΕ. Όσο περισσότερες φιλοδοξίες έχουμε για τη μείωση των εκπομπών, τόσο πιο σημαντικό και απαραίτητο γίνεται ιδιαίτερα στις περιφέρειες όπως είναι η βυρική Χερσόνησο, εκεί που έχουμε σαφές έλλειμμα και πρόβλημα διασύνδεσης. Ε, είπε ο Κλωτούρμες ότι θα γίνουμε ε, καθαρή εξαγωγή. Όχι, δεν θα, θα μπορέσουμε να εξάγουμε τίποτα, γιατί δεν θα μπορέσουμε να αυξήσουμε την παραγωγή μας μέσω ΑΠΕ αν δεν θα έχουμε διέξοδο. Οπότε Θέλουμε μέσο και μακροπρόθεσμη προοπτική και μέσο μακροπρόθεσμο ορίζοντα για όλα τα σχέδια και τις αποφάσεις κοινού ενδιαφέροντος. Δεν μπορούμε να είμαστε μόνο κοντόφθολμοι και βραχυπρόθεσμοι. Δεν θα έχουμε έτσι το πραγματικό ε, ενδιαφέρον ε, και συμφέρον για ένα σχέδιο κοινού ενδιαφέροντος, αν δεν υιοθετήσουμε μια πιο μακροπρόθεσμη προοπτική. Σας ευχαριστούμε κυρία Πιλάρτα Τελκαστήγιο. Τώρα κύριε Γενική Διευθυντά, Έχετε το λόγο εσείς, γιατί ακούσετε όλες τις παρατηρήσεις και όλη την υποστήριξη από την Επιτροπή, αλλά και πολλές απορίες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ σε όλους για τα σχόλιά σας και την υποστήριξη που μου προσφέρετε. Απευθυνόμενος στον εισηγητή, θέλω να πω ότι αναμφισβήτητα ε, θα γύρουμε γέφυρες ε, ανάμεσα στα διάφορα στοιχεία που αφορούν στο μηχανισμό συνδέοντα στην Ευρώπη. Ενέργεια, μεταφορές, ψηφιακό κομμάτι, όλα αυτά προφανώς και εντάσσονται μέσα στη διαδικασία εξυγχρονισμού. Και πρέπει ε, να προτείνουμε και εναλλακτικέ λύσει. Ήδη υπάρχει ένα πρόγραμμα όπου συμμετέχουν η Γαλλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίση, ε, θα δώσουμε τη δυνατότητα να υπάρχουν ε, ε, διατομεακές συνέργειες. Ε, ως προς την ψηφιοποίηση. Αυτή θα είναι απολύτως απαραίτητη κατά τα επόμενα έτη. Ε, για μεγάλο χρονικό διάστημα υπήρχε αντίδραση να ακολουθήσουμε αυτή την κατεύθυνση. Τώρα όμως αυτό είναι απολύτως απαραίτητο όχι μόνο για να βελτιωθεί η απόφαση των δικτύων, αλλά και για να υπάρχει και για μεγαλύτερη ασφάλεια, για να μπορούμε παρά αυτά να εντοπίσουμε κάποιο ατύχημα που μπορεί να συμβεί στο δίκτυο και να επεμβαίνουμε με μεγαλύτερη ταχύτητα. Το ίδιο ισχύει και για την κυβερνοασφάλεια. Ε, οι υποδομές, κρίσιμες κυρίως αυτές τις ενέργειες, είναι ένα καθοριστικό στοιχείο της ε, κυβερνοασφάλειας. Πέρα από όλα αυτά πρέπει να υπάρχει σχέση ανάμεσα στην ενέργεια, τις μεταφορές, το ψηφιακό κομμάτι, αλλά και τα διαρθρωτικά ταμεία και το πρόγραμμα ορίζοντας για την Ευρώπη. Όσον αφορά τη δεύτερη παρατήρηση από τη συνάδελφο, η ε, ηλεκτρική ενέργεια πράγματι θα καταστεί η πραγματική προτεραιότητα ε, και θέλω να σας πω, επειδή πολλοί από εσάς ε, αναφερθήκατε σε αυτό το θέμα, θα ήθελα λοιπόν να σας πω ότι η άποψή μου είναι ότι θα πρέπει να φτάσουμε στο τουλάχιστον 85 με 90% ε, προγράμματα ηλεκτρικούς, ηλεκτρικής ενέργειας ε, στο νέο πολιετές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο, να χρηματοδοτούνται δηλαδή αυτά. Γιατί θεωρώ ότι όλα αυτά είναι απαραίτητα. Το νέα πήγαμε στη Σόφια και την Πρατισλάβα και είδαμε τραγική η κατάσταση Αυτές οι χώρες κατά 100% εξαρτώνται από το αέριο της Ρωσίας. Μετά την κρίση Ρωσίας-Ουκρανίας υπήρξε διατραχή στον εφοδιασμό και αυτό ήταν καταστροφικό όχι μόνο για οικονομικούς λόγους, γιατί δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν ε, τα εργοστάσια, αλλά και για τους πολίτες, ε, τα νοσοκομεία, τα σχολεία, δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν. Ως εκ τούτου, ε, θεωρούμε ότι είναι απολύτως απαραίτητο να ακολουθήσουμε πρώτα απ' όλα αυτή την κατεύθυνση και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Κοινοβούλιο για την ε, ταχύτατη ολοκλήρωση του κανονισμού περί αερίου. Αυτό είναι ένα καθοριστικό στοιχείο όλων αυτών των θεμάτων που αφορούν σε ασφάλεια. Κατά τα άλλα, να σας πω ότι θα αποδώσουμε ιδιαίτερη σημασία στη νέα υποδομή για το αέριο, κυρίως στον αγωγό της Βαλτικής από την Ορβηγία, Δανία, στην Πολωνία. Πολύ σημαντικός αγωγός αυτός, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, ε, στο πλαίσιο της διαφοροποίησης της χώρας σας ε, ενεργειακά. Τα πράγματα προχωράνε πολύ καλά, θα έλεγα, και αυτά κατ' ουσίαν σημαίνουν και άλλη μία επιτυχία προς την κατεύθυνση της διαφοροποίησης, ενεργειακής διαφοροποίησης. Συμφωνώ μαζί σας με τη σκέψη σας όσον αφορά την κινητικότητα με βάση την ηλεκτρική ενέργεια. Πολλά κρατημέλη ε, ανθίστανται στο να διευκολύνουν την ανάπτυξη σημείων ε, φόρτισης ε, σε εμπορικούς χώρους, σε επαγγελματικούς χώρους, κυρίως στις αστικές περιοχές, όπου έχουμε υψηλό επίπεδο ρήπανσης. Και όπως πολύ καλά γνωρίζετε, θέλουμε να επιταχύνουμε σε αυτή τη νέα κατεύθυνση. Εξάλλου, θα αποδώσουμε ιδιαίτερη σημασία σε όλα τα θέματα της ε, διαλειτουργικότητας, της διασύνδεσης, των δικτύων. Προς τον κύριο Μόρταν θέλω να πω ότι πρέπει να αυξήσουμε τη συμβολή του Συνέδρου στην Ευρώπη στη μείωση των εκπομπών. Γνωρίζετε όμως πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή Για να μειωθούν οι εκπομπές πρέπει να συνδυαστεί η καθαρή ενέργεια, κυρίως η ΑΠΕ, και με την ενεργειακή απόδοση και με την διασύνδεση των δικτύων. Αναφορθήκατε στη μακροχρόνια κατάργηση του άνθρακα, στα νέα κριτήρια. Ε, πράγματι πρέπει να διασφαλίσουμε ότι για αυτή τη μεταρρύθμιση ε, δεν θα καταλήξουμε στο λιγότερο από 85-90% προτεραιότητα στην ηλεκτρική ενέργεια. Και είμαι σίγουρος ότι έχουμε τη δυνατότητα να το καταφέρουμε αυτό. Η Ευρώπη θα ηγείται στον κόσμο Ελπίζω με ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο, αλλά και με τη δυνατότητα να μετακινηθεί απολύτως προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν βλέπω να υπάρχει άλλος ανταγωνιστής στον κόσμο που να φτάνει ε, στο 50% χρήση των ΑΠΕ κατά τα επόμενα 10 χρόνια. Και κύριε Μπλανκολόπης, εμείς νομίζω μπορούμε να ξεπεράσουμε και το 50% μπορούμε να το ξεπεράσουμε το 50% γιατί δημιουργούμε μια, ένα δυναμισμό και όπως ξέρετε ο τελευταίος ε, τριμής διάλογος ολοκληρώθηκε με στόχο τουλάχιστον 32%. Και με το, την προοπτική της αναθεώρησης. Νομίζω λοιπόν ότι ε, ήταν πολύ καλές αυτές οι διαπραγματεύσεις. Κύριε Μαρτσελέζη. Θα σας έλεγα ότι όντως στην αρχή χρειάστηκε να ασχοληθούμε με το φυσικό αέριο, λόγω της εξαιρετικά δύσκολης κατάστασης που αντιμετωπίζαμε σε πολλά τμήματα της Ευρώπης και κυρίως στη κεντρική και ανατολική Ευρώπη και στη νότιο ανατολική Ευρώπη. Και σημειώσαμε τεράστια πρόοδο έκτοτε. Στόχος μας είναι μέχρι το 2020 να μην υπάρχει ούτε μία χώρα που να εξαρτάται απολύτως από έναν και μόνο προμηθευτή. Και ήδη μπορούμε τώρα να δώσουμε την απόλυτη προτεραιότητα στην ηλεκτροδότηση, στην ηλεκτρική ενέργεια και ανταποκρινόμενοι στο αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ανοίξουμε ένα νέο παράθυρο στο ΣΕΦ για τις ΑΠΕ, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ό,τι αφορά την Ιβηρική Χερσόνησο και εκεί έχουμε μια πολύ σημαντική ευκαιρία και με το Βασκονικό κόλπο γιατί έχουμε πια τρεις χώρες ε, για τις ε, διασυνδέσεις μεταξύ των τρίτων χώρων. Το σχέδιο αυτό για το Βασκονικό κόλπο είναι πολύ σημαντικό και έχει ένα μεγάλο τμήμα ε, στη θάλασσα και μάλιστα αυτή τη στιγμή ε, εργαζόμαστε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πολύ έντονα στηρίζοντας πρωτοβουλίες που θα λάβουν την τα δημόσια, δημόσια υποστήριξη για δημόσια κονδύλια. Για παράδειγμα, υπάρχει η πρωτοβουλία για τα ανανεώσιμα δίκτυα που γίνεται σε συνεργασία με τους διαχειριστές δικτύου, πολλούς διαχειριστές δικτύου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και με πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις, προκειμένου να αποδείξουμε στο κοινό, στον κόσμο, τι ωφέλη μπορεί να αντλήσει από την προσέγγιση αυτή. Οφέλη και ως προς την ασφάλεια, αλλά και ως προς την ανταγωνιστικότητα των τιμών, αλλά και ως προς την διάρκεια και τη βιωσιμότητα. Και είναι πολύ σημαντικό να αναβαθμίσουμε τις δράσεις μας στο τομέα αυτό. Και πιστεύω ότι στις ε, τελικές διαπραγματεύσεις που θα έχουμε για το θέμα αυτό, να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση σε αυτό το θέμα. Θα αναθεωρήσουμε τα κριτήρια. Αλλά αν καταφέρουμε να δώσουμε προτεραιότητα σε αυτά τα θέματα. ηλεκτροδότηση, αλλά και διασυνοριακά σχέδια μίζωνος σημασίας, με βάση την περιφερειακή εμπειρία που είχαμε και που είναι πολύ καλή παντού στην Ευρώπη, πιστεύω θα έχουμε κάνει το σημαντικότερο βήμα. Για την κυρία Βέρνερ, θα ήθελα να πω ότι 10 κράτη-μέλη και όχι από τα μικρότερα, βρίσκονται κάτω από το 10% διασύνδεση, οπότε θα πρέπει να συσπυρώσουμε τις προσπάθειές μας και τις δράσεις μας. Έχουμε και μια ομάδα υψηλού επίπεδου που λειτουργεί πολύ καλά και μαζί με αυτή την ομάδα έχουμε το στόχο του 15% στη διασύνδεση και πιστεύω ότι θα έχουμε τα μέσα να εφαρμόσουμε αποτελεσματικές παραμέτρους με ανάμειξη όλων των ε, παραγόντων και τις ρυθμιστικές αρχές και τα κράτη-μέλη και τους TSO, τους διαχειριστές ε, δικτύων με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και κυρία Γκροστές, ο, Γκροστέτ, όντως η αποδοτικότητα είναι από τα κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη για την ε, επιλογή των σχέδιων. Δεν θα είναι όμως το μόνο κριτήριο η αποδοτικότητα αλλά έχουμε ένα σύστημα επιλογής ε, που είναι καλά ρονταρισμένο και έχει ως πρωταρχικό άξονα τις περιφέρειες και ε, ε, προσελκύει και τα κράτη-μέλη και αναμειγνύει τα κράτη-μέλη και τους DSO και έχουμε μια κατανομή του κόστους σε συνεργασία με τις, τις ρυθμιστικές αρχές. Πάντως, η μεσοπρόθεσμη χρηματοδότηση για τα ενεργειακά προγράμματα υπερβαίνει κατά πολύ την αντίστοιχη χρηματοδότηση στον τομέα των μεταφορών, για παράδειγμα. Και έχουμε και αυξημένη ανταγωνιστικότητα σε ολόκληρη την ενεργειακή αλυσίδα, ακόμη και για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κάτι που δεν ίσχυε μέχρι σχετικά πρόσφατα. Έτσι έχουμε επιπλέον επιχειρήματα για να οδεύσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Κύριε Μπλάνκο Λόπες, όντως αυτό είναι ένα απαραίτητο στοιχείο αυτό της διασύνδεσης στο γενικό θέμα της Ενεργειακής Ένωσης. Και μάλιστα το έργο σας ως συγητού για τη ΣΑΠΕ ήταν ε, πραγματικά πάρα πολύ αξιόλογο και αξιέπαινο και είχαμε πολύ ε, επικοδομητική συνεργασία με την Προεδρία, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη-μέλη αλλά και όλους τους ενδιαφερόμενους. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να έχουμε αγαστή συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Και σίγουρα ο ρόλο τη διασύνδεση σε συνδυασμό με τι ανανεώσιμε πηγές ενέργεια είναι τεράστιο. και ήταν από τι σημαντικότερε προκλήσεις που είχαμε να αντιμετωπίσουμε, αλλά και από τι μελλοντικέ προκλήσει. Αλλά είναι πολύ θετική αυτή η πρόκληση. Είπα στον κύριο Μαρτά ποια ήταν η γνώμη μου για τι περιφέρειες και αυτό ισχύει και για την COP24. Πιστεύω ότι χάρη στη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και με το Συμβούλιο θα φτάσουμε στην COP24 στο Κατοβίτσα με, με την καλύτερη προετοιμασία. Και αυτή η καλή προεργασία και προετοιμασία θα αυξήσει τις διαπραγματευτικές μας ικανότητες, κυρίως για την ηλεκτρική ενέργεια και για την καλύτερη αξιοποίηση του τεράστιου δυναμικού της αγοράς. Σήμερα το ψηφιακό, ο ψηφιακός τομέας είναι στις αναπτυσσόμενες χώρες ε, το 15-16% της, κατανάλωσης, της ενεργειακής κατανάλωσης. Το ίδιο ισχύει και με την ηλεκτροκίνηση. Και εκεί θα α, χρειαστεί αύξηση της παραγωγής, αλλά με γνώμονα και την ποιότητα. Και από αυτή την άποψη πιστεύω ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Κλοντ Τούρμες, συμφωνώ απόλυτα με την ανάλυση σας και τα λεγόμενα σας. Σίγουρα θα πρέπει ε, να προετοιμαστούμε πολύ καλά στη διαπραγμάτευση με το Συμβούλιο, να έχουμε καλά και πιστικά επιχειρήματα και νομίζω ότι αδειάστητα επιχειρήματα έχουμε με το επίπεδο ανταγωνιστικότητας και το δυναμικό της αγοράς που είναι ορατό παντού στην Ευρώπη, όχι μόνο στη Βαλτική αλλά και αλλού. Και είχαμε πολλές καλές ε, συζητήσει ε, και στο Κατοβίτσε που ήταν πολύ ενθαρρυντικές και τώρα βλέπουμε την Πολωνία να βγάζει σε πληστηριασμό χιλιάδες μεγαβάτ και μάλιστα να υιοθετεί, να υιοθετεί πολύ πιο θετική εθνική νομοθεσία. Αλλά τέτοιου είδου δράσεις και στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη αλλά και αλλού και στην Νότιο Ανατολική Ευρώπη αλλά και στην Νοτιοδυτική Ευρώπη και στην Κεντρική Ευρώπη είναι πολύ σημαντικές ενέργειες ώστε τι θετικέ περιφερειακές εμπειρίες να τις αξιοποιήσουμε για να δημιουργήσουμε ανταγωνιστικές και ευρύτερε αγορές. Και συμφωνώ επίσης ε, με το σχόλιο σα για τη βιομηχανική βάση και το σχόλιο της κυρίας Δελκαστήγιο για την ε, ταυτόχρονη ανάπτυξη των διασυνδέσεων και την τήρηση των στόχων. Γιατί αν δεν δώσουμε έμφαση και στην διασύνδεση και στου στόχου δεν θα καταφέρουμε να υλοποιήσουμε όλου του κοινού μα στόχου. Και νομίζω ότι σήμερα έχουμε πολύ περισσότερα του στη διάθεσή μα για να υλοποιήσουμε του στόχου μα. Και τέλο ήθελα να πω ότι οι διασυνδέσει μα φέρνουν πιο κοντά. Φέρνουν πιο κοντά όχι μόνο τι αγορέ, αλλά και τι χώρε και τον πληθυσμό των χωρών. Και γι' αυτό έχει νόημα εκείνη η προσπάθεια προς την ενίσχυση της διασύνδεσης. Ευχαριστώ. Εμεί ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος, κύριε Γενική Έγνα Και... Η συνεργασία της Γενικής διευθυντή σας υπό τη δική σας διοίκηση συνεργάζεται πάρα πολύ με την ε, Επιτροπή μας και σας διαβεβαιώ όπως ανέφερε η κυρία Συγήτρια ότι εμείς θα κάνουμε ό,τι πέρα από το χέρι μας, ούτως ώστε να εγκριθεί αυτή η σημαντική πρόταση που αποτελεί η αρμοδιότητά μας. Και πάλι ευχαριστούμε. Thank you. Yeah, thank you very much. Uh, dear friends, uh, Πάμε, συνάδελφοι, τώρα στο τελευταίο θέμα, για το οποίο δεν έχουμε πολύ χρόνο για την ενημέρωση όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις. Είναι το τελευταίο μας θέμα πριν τη μεσημερινή διακοπή. Είναι το σημείο υπερδημών 17. Εδώ έχουμε δύο πολύ σημαντικές ε, εκθέσεις. Αφορούν την ψηφιακή Ένωση. Η ψηφική ένωση είναι η αρμοδιότητά μας και πριν από δύο εβδομάδες με επιτυχία ολοκληρώσαμε δύο σημαντικές νομοθετικές προτάσεις. Πρώτα-πρώτα τον κώδικα για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες της Ευρώπης και επίσης την έκθεση για τους ε, αρμόδιους για αυτό το θέμα ε, ρυθμιστικούς οργανισμούς. Έχουμε τώρα την κυρία Πιλαρδέλ Καστίγιο, που είναι μία από τους ε, εισηγητές, ως αφορά κώδικα των ηλεκτρονικών ε, επικοινωνιών, και από την άλλη έχουμε τον κύριο Εύζεν Τοσενόφσκι, που είναι ο άλλος συνεισηγητής. Πέστε μας. Πώς πάνε οι διαπραγματεύσεις. Είναι πολύ καλό το αποτέλεσμα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να σας τα πω πιο γρήγορα και στα αγγλικά και στη μητρική μου γλώσσα. Όχι, θα πω στη μητρική μου γλώσσα καλύτερα από πλευράς των θέσεων του Κοινοβουλίου η συμφωνία που αποσπάσαμε πριν από δύο εβδομάδες ήταν μια επιτυχία. Ήταν συμφωνία με το Συμβούλιο. Και ε, αυτή η πρόταση είχε στόχο να είμαστε υπέρ κάποιες ρυθμιστικής αρχής που να μας δίνει το πιο προβλέψιμο. Να περιορίζονται οι κίνδυνοι και έτσι να έχουμε δίκτυα υψηλών δυνατοτήτων. Και έτσι να φτάσουμε σε ένα επίπεδο συνδεσιμότητας που ακόμα δεν το έχουμε πετύχει, αλλά έχουμε κάποιες προβλέψεις ε, της Επιτροπής που θα έχουμε οδηγήσει σε επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα 500-600 δισεκατομμυρίων. Επομένως ε, ε, πρόκειται για κάτι που είναι στην καρδιά αυτής της νομοθεσίας και γι' αυτό και έχουμε επίσης προστα... την προστασία των καταλωτών ως αρμοδιότητα και επίσης της ενιαίας αγοράς. Πάντως, αναβαθμίζεται τώρα αυτή η υπόθεση της ε, αγοράς στα πλαίσια αυτής της ε, νομοθεσίας παραδείγματα μέτρων πρώτα-πρώτα τήρηση που προβλέπονται για το ε, ραδιοελεκτρικό φάσμα και όσον αφορά την διαχείριση δεν υπήρχε καμία εναρμόνιση, δεν είναι εθνική αρμοδιότητα αποκλειστικά. Τώρα έχουμε όλα αυτά τα μέτρα τα οποία αφορούν ε, και τις αδειοδοτήσεις της 20 ετής και επίσης ε, παρέχεται η εγγύηση ότι δεν θα έχουμε στις αναθέσεις κάποιες ε, αλλαγές, ότι θα υπάρχει διαφάνεια, θα υπάρχει δικαίωμα σε αποζημίωση για τις σχετικές εγκρίσεις άδειες όταν έχουμε κάποια μισθώματα και είπαμε ότι θα πρέπει τα κρατημέλη να απορριθμίσουν την αγορά όσον αφορά το 5G και αυτά πριν το 2020 ούτως ώστε να έχουμε τέτοιες συνθήκες στην Ευρώπη για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε την τεχνολογία πέμπτης γενιάς 5G. Τώρα όσον αφορά την αντιστάθμιση του κινδύνου, το νέο πρότυπο που ε, θεσπίζεται είναι η αποκοινού επένδυση που θα αφορά αυτά τα νέα δίκτυα, τα οποία θεσπίζονται και οι ρυθμιστικές αρχές θα μπορούν να έχουν την κριτική ευκαιρία για το τι συμμετοχή θα υπάρχει όταν πληρούνται κάποιε προϋποθέσεις και θα υπάρχει αντισταθμίση κινδύνου γιατί έτσι θα υπάρχει περισσότερη ασφάλεια, βεβαιότητα που ευνοεί τις επενδύσεις. Και με αυτή την απόφαση καλύπτουμε τώρα τις διεθνείς κλήσεις, calls» όπως τις λέμε, και τώρα το κόστος είναι 19 λεπτά το λεπτό. Τώρα είναι 19. πάμε για 45. Η 45 είναι και θα φτηνίνει στα 19, ούτως ώστε να έχουμε όταν έχουμε κάποιο είδους χονδρική πώληση, πάμε στα 3,5. Μέχρι 65 φτάνει σε κάποια χώρα. Οπότε τώρα έτσι πλησιώσαμε την πρόταση της Κομισιόν. για τη ρύθμιση της ε, αγοράς των τηλεπικοινωνιών. Τα δεδομένα, η περιαγωγή, αυτά προσέξαμε που είναι σημαντικά και αυτά καλύψαμε με αυτή την ε, νομοθεσία. και να ευχαριστήσω όλους τους κοιοδησηγητές και όλους που μας βοήθησαν. Ήταν πάρα πολύ καλή η συνεργασία μας με την γραμματεία και μας βοήθησε για το θέμα. Ο Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Τώρα για, το, για την, τον οργανισμό Μπέρεκ, ο κύριος Πασενόφσκι. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ε, εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς την κυρία Πιλάρ Καστίγιο για την προσπάθεια που έκανε και το πολύ αξιόλογο έργο της για τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Ελεκτρονικών Επικοινωνιών. Πετύχαμε όσα ζητούσαμε και κυρίως να συντονιστούμε στις δύο εκθέσεις για τον ΠΕΡΕΚ, τον Ευρωπαϊκό Φορέα Αριθμιστικών Αρχών για τις Ελεκτρονικές Επικοινωνίες και, το... και τη δική της έκθεση για τον ε, κώδικα. Και μάλιστα είναι ενδεικτικό ότι την ίδια μέρα, μάλλον την ίδια νύχτα, ολοκληρώθηκαν οι αντίστοιχοι τριμερεί διάλογοι. Και ευχαριστώ θερμά την κυρία Καστίγιο για τη συνεργασία που είχαμε. Ήταν πολύ δύσκολο να καταλήξουμε σε συμβαστική λύση και αντιλαμβάνομαι ότι δεν έμειναν όλοι πλήρω ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα, αλλά σε περίπλοκες εκθέσει ε, είναι αναμενόμενο κάτι τέτοιο. Και μάλιστα το Κοινοβούλιο ήταν διχασμένο αρχικά ω προ την ε, ίδρυση ενός οργανισμού με τη συγχώνευση του Μπερέκ και του γραφείου Μπερέκ. Τελικά καταφέραμε να ξεπεράσουμε τη δυσκολία και ε, να καταλήξουμε σε μια δεσμευτική απόφαση διαφυλάσσοντας το δετό χαρακτήρα της δομής του Μπερέκ που ήταν και η κατάλληλη λύση αυτή τη στιγμή. Πιστεύω ότι σύντο χρόνο θα γίνουν πολλές αλλαγές και εξελίξεις στην αγορά τηλεπικοινωνιών και θα αυξηθούν και οι προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει ο Ευρωπαϊκός Φορέας Ρυθμιστικών Αρχών για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, ο Μπερέκ. Γι' αυτό και πιστεύω θα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί ως προς τις αλλαγές και να τις αγκαλιάσουμε. Και μετά από λίγο καιρό θα χρειαστεί να αναθεωρήσουμε και το μοντέλο που υιοθετήσαμε μέχρι τώρα. Θα πρέπει να, πρέπει να είμαστε πάντως διαλλακτικοί και ανοιχτοί ω προ τι πιθανές αλλαγές. Ευχαριστώ τους και οδησηγητές, τους συναδέλφους, τη γραμματεία, γιατί πραγματικά ήταν σημαντική αρρωγή της σε αυτή την περίπλοκη διαπραγματευτική διαδικασία. Προσπαθήσαμε να συσπηρωθούμε για να περάσουν ε, τα επιχειρήματά μας και οι απόψεις μας. Ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υποστήριξή της, την Επιτροπή μας μάλλον, την Επιτροπή Ήτρε και τους εμπειρογνώμονές μας που μας βοήθησαν πολύ και καταλήξαμε να διεκπαιρώσουμε αισίως τον τριμερή διάλογο για τον Μπερέκ. Λύσαμε και τα προβλήματα με τους κανόνες για τη δικαιώματα ψήφου. Οπότε είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος για το ότι ολοκληρώσαμε τον τριμερή διάλογο με λογικό αποτέλεσμα και κυρίως ε, διεκπαιρώσαμε ένα τόσο σημαντικό θέμα. Ναι, και για τις δύο περιπτώσεις ε, είχαμε παράλληλες διαπραγματεύσεις, οπότε θα ζητήσουμε από εκείνο τα δύο θέματα. Η κυρία Νίμπλερ, ο κύριος Σον δεν ξέρω άλλος κανείς θέλει το λόγο. Όχι, κυρία Νίμπλερ και μετά ο Σον Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δράτομαι και εγώ τις ευκαιρίες ε, να ευχαριστώ την εισηγητριά μας, την κυρία Ντεκαστήγιο, όπως επίσης ε, και τις ε, άλλες συναδέλφους. Σας ευχαριστώ όλους θερμά. Πραγματικά προέκυψε ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα και ο συνάδελφος, ο προαλήσεως, ο κύριος Τισανόσκη, το είπε ήδη ότι εδώ στο Κοινοβούλιο είναι πολύ δύσκολο να επιτύχει κανείς μια κοινή γραμμή και μετά να την περάσει και στα κράτη-μέλη. Αυτό το θέμα για μένα είναι σημαντικό. Το είπε και η συγγήτρια. Οφείλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα γίνουν επενδύσεις ε, στην υποδομή των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Μιλάμε για δισεκατομμύρια τα οποία πρέπει να επενδυθούν και γι' αυτό λοιπόν αν δεν δημιουργήσουμε κίνητρα για την ευρωπαϊκή αγορά για να γίνουν επενδύσεις στην υποδομή των ηλεκτρονικών επικοινωνιών τότε αυτό θα σημαίνει ότι δεν κάναμε καλή δουλειά. Ελπίζω λοιπόν με τη συμβαστική πρόταση να έχουμε πετύχει κάποια ισορροπία. Δηλαδή να έχουμε έτσι ώστε τα συμφέροντα των ε, καθιερωμένων παρόχων να λαμβάνουν υπόψη, αλλά να μην αγνοούνται και οι μικρές επιχειρήσεις που θέλουν και αυτές να μπουν στην αγορά. Να έχουν και αυτές αυτή τη δυνατότητα. Για τους ε, πολίτες μας θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό ε, στα, στους ενδοευρωπαϊκούς διαγωνισμούς να γίνεται ένα βήμα προς τα εμπρός. Εμείς ως Κοινοβούλιο είμαστε υπέρ της ε, κατάρρησης περιαγωγής. Είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να τηλεφωνούμε χωρίς να καταβάλουμε συνεισφορές. Ε, πραγματικά αυτό είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία ξεκίνησε από το Κοινοβούλιο και σήμερα νομίζω ότι θα πρέπει κανείς να το επαναφέρει στη μνήμη μας. Ευχαριστούμε όλους που βοήθησαν στο να επιτευχθεί αυτό το τόσο σημαντικό αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ καταρχήν την Πιλάρ για την πολύ καλή δουλειά της. Ευχαριστώ και τους Σκιώτης γιατί το αποτέλεσμα σε γενικές γραμμές ε, είναι πολύ ικανοποιητικό. Εγώ είμαι ευχαριστημένη και άλλοι είναι ευχαριστημένοι. Ε, το είπε και η Αγγέλικα. Ε, οι μακροχρόνιοι πάροχοι μπορούν να παραμείνουν στην αγορά, δεν εκδιώκονται, αλλά ακόμα πιο σημαντικό λαμβάνεται υπόψη ο καταναλωτής. Ο συμβασμός ήταν απαραίτητος, γιατί έτσι οι πάροχοι κατ' ουσίαν δεν μπορούν πια να αυξάνουν ε, κατά τις ε, τιμές ε, για να προσπορίζονται περισσότερα κέρδη. Γι' αυτό είχε ξεκινήσει καταρχήν και η κατάργηση της περιεγωγής. Αυτό είναι μια πολύ καλή έκθεση, μας αρέσει πολύ και άλλη μια φορά δείχνει το Κοινοβούλιο οι βουλευτές μπορούν να λάβουν υπόψη τους τα συμφέροντα των πολιτών και αν δεν το κάνουν οι πολίτες ε, οργίζονται, ψώνουν τη φωνή τους. Πιλάρ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά που έκανες. Σε ευχαριστούμε και τους ε, συναδέλφους. Πρόεδρος, ε, να πω ε, το ίδιο θα πω πάλι και στους δυο σας απευθυνόμενους. Πραγματικά, συνάδελφοι, τα καταφέρατε καταπληκτικά. Συγχαρητήρια, ε, συγχαρητήρια για την πολύ καλή δουλειά σας, γιατί δεν είναι εύκολο να πετύχει κανείς ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Αν λοιπόν θέλουμε να αισθανόμαστε ως Επιτροπή ότι επιδεικνύουμε υπευθυνότητα, θα πρέπει συνεχώς και στο μέλλον να προβάλλουμε τέτοιου είδους ε, λύσεις. Πολύ καλό το ότι μπορέσαμε αυτή τη φορά να παρουσιάσουμε αυτό το αποτέλεσμα. Είμαστε ανοιχτοί και μπορούμε και να συζητάμε, ακόμα και αν υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, διαφορετικές πολιτικές θέσεις ως πολιτικές ομάδες. Ευχαριστούμε πολύ για την ε, υπομονή σας. Ε, και θέλω να πιστεύω ότι θα μπορέσετε να αντέξετε και σήμερα το βράδυ μέχρι και αργά το πρωί γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό ε, να παρουσιάσετε στους πολίτες ε, κάτι που να είναι χειροπιαστό. Ευχαριστούμε βεβαίως και τους σκιώδης ηγητές γιατί χωρίς σκιώδης ηγητές δεν θα ήταν δυνατόν να έχουμε επιτύχει αυτό το εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Ψηφιακή Ευρώπη λοιπόν. Βεβαίως υπάρχει μπροστά μας η Ενεργειακή Ένωση. Ποτέ δεν τελειώνει η δουλειά, υπάρχουν και θέματα του προϋπολογισμού, εν πάση περιπτώσει. Πολύ ωραία. Προχωράμε τώρα στην Ενεργειακή Ένωση. Και Έχουμε τον συνάδελφο κύριο Πόχα, ο οποίος είπε, μίλησε προηγουμένως πριν από μία ώρα, τώρα προαγωγή της χρήσης ενέργειας από τη ΣΑΠΕ. Αναδιατύπωση Συνάδελφος Χωσέ Μπλανκολόπης. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ με την ευκαιρία να συγχαρώ την Πιλάρ, διότι ήταν το έργο της πάρα πολύ αξιόλογο, ενώ είχε λίγο χρόνο και ήταν και δύσκολα. Και εμείς ε, τα, τα στις 13 του καταφέραμε να κλείσουμε αυτή τη συμφωνία για αυτή την οδηγία που είναι πολύ σημαντική για τις ανανεώσιμες ενέργειες 2020-2030. Πρώτα-πρώτα να ευχαριστήσω τους κοιόδες εισηγητές, κάποιοι από αυτούς είναι εδώ, κάποιοι λείπουν, ο κύριος ε, Κέλλη, ο κύριος ε, Τούρμες, όλους, όλους να ευχαριστήσω που μας βοήθησαν ε, και έτσι καταφέραμε να έχουμε επιτυχή κατάληξη. Υπάρχει τώρα το 32% δεσμευτικό στόχο για όλη την Ευρώπη με ορόσημο το 2030 και ξεκίνησαμε το 27% που ήταν η πρόταση του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και είπαμε αυτό το 2023 επιδέχεται μια αναθεώρηση προς τα πάνω για τη εξέλιξη των δαπανών του κόστους. Εάν συνεχιστεί η τωρινή τάση, πρόκειται να μας επιτρέψει να πάμε ακόμα παραπέρα όσον αφορά τη φιλοξευτή συμφωνία. Επίσης, έχουμε κάποιους τομείς που καταλώνουν πολύ ενέργεια, εκεί θα πρέπει να μπουν τα ανανεώσιμα στην ψήξη, στη θέρμανση και βέβαια όσον αφορά τις μεταφορές με το στόχο του 14% που και αυτό επιδέχεται θεώρησε το 23%. Επίσης όσον αφορά τις συγκρίσεις, τις, ε, ε τις συγκρίσεις για τα ε, καύσιμο πρώτης γενιάς, παγώνουν αυτά για κάθε κράτος το 20. Ακριβώς όπως έχει εγκρίνει το Κοινοβούλιο. Σε καμία περίπτωση είναι δυνατόν να ξεπεράσουμε το 7%. Οπότε αυτά όλα μπήκαν εδώ όσον αφορά μεταφορές και αυτό είναι διακριτική ευκαιρία των κρατών και όσον αφορά τώρα τα προχωρημένα έχουμε ένα 3,5% για το 2030 αυτές τις προοδευτικές τους και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα βίο τα προχωρημένα. Κάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ διαφορετικό στο κοινοβούλιο ήταν τα σχετικά με το φινικέλαιο και εδώ ήταν πάρα πολύ θετική συμφωνία ε, γιατί είπαμε να υπάρχει κατάργηση των δύο ε, καυσίμων της βιομάζας ε, που έρχονται από κάποιες ε, καλλιέργειες. Εκεί που προβλέπεται να υπάρξει επέκταση της καλλιέργειας, εκεί όπου υπάρχει θέμα από θέματος διοξιδίου. Το 2019 παγώνει και από το 2023 η συμβολή θα αρχίσει να συρρυκνώνεται, ούτως ώστε να φτάσει το 0% το 30% η Επιτροπή με τη πράξη πρόκειται να καθορίσει τα κριτήρια για την πιστοποίηση για αυτά τα βιοκαύσιμα όπου είναι μικρό ο κίνδυνος αλλαγής της χρήσης της γη. ό,τι στοιχεία υπάρχουν και επίσης με στην πράξη θα ορίσει το πώς θα γίνει η βαθμιαία ε, σύρρυκνωση, μείωση της χρήσης αυτών των βιοκαυσίμων. Επίσης, όσον αφορά την αυτοκατανάλωση εδώ υπήρχε θέμα ερμηνείας, ξεκαθαρίστηκε, αφορούσε κάποια ημερομηνία και όπως γνωρίζετε για μένα είναι σημαντικό. Όπως και να έχει, κατοχυρώνεται το δικαίωμα στην αυτοκατανάλωση για να να, να παράγει, να αποθηκεύει και να καταναλώνει. Επίσης κατοχυρώνεται για όταν υπάρχει κάποιο πλεόνασμα το οποίο πηγαίνει στο δίκτυο, στην τιμή της αγοράς. Επίσης, καθιόνται η αρχή του να μην υπάρχουν κάποιες ε, χρεώσεις. Και αυτό θα είναι γενικός κανόνας με κάποιες εξαιρέσεις σε κάποιες περιπτώσεις. Είναι κατακλείδη, ήταν πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα οποία αποσπάσαμε τελευταίο 1,5 χρόνο, οπότε σήμερα είμαστε σε θέση να πανηγυρίσουμε για αυτή τη συμφωνία που πετύχαμε και βέβαια επέδειξε καλή θέληση το Συμβούλιο όσοι ε, συνεργάστηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υπήρξε προσπάθεια ιδιαίτερη που καταβάλαμε ούτω ώστε να καταλήξει το Κοινοβούλιο σε μια ομόφωνη τοποθέτηση σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Ομοφώνησαν όλες τις πολιτικές ομάδες και αυτό είναι και τη θέση μας. Νίμπλε. Oh, well, sorry, uh, shadow reporter. Okay, of, Συγγνώμη πρώτα και ο Ναι, βεβαίω. Βλέπω ότι κοιτάτε το ρολόι, οπότε θα είμαι σύντομος. Πραγματικά ήταν μεγάλη τιμή που συμμετείχα σε αυτές τις συζητήσεις. Ε, πολύ δύσκολο θέμα, εξαιρετικά περίπλοκο. Είχαμε πολλές δυσκολίες για τα βιοκαύσιμα για πολύ καιρό. Τελικά καταλήξαμε σε ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα και μπράβο στον εισηγητή μας, τον κύριο Μπλάνκο Λόπες, που ήταν πολύ διαλλακτικός, ε, είχε μεγάλη κατανόηση και φρόντισε να διασφαλίσει την αυτοκατανάλωση και να της δώσει προτεραιότητα. Τα κατάφερε. Συγχαρητήρια. Και ευχαριστώ και τον πρόεδρο Μπούζεκ που προείδευσε ε, στους τριμερείς διαλόγους. Το τελευταίο κράτησε 10 ώρες με, από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 4 τα χαράματα. Αλλά ήταν πολύ θετικό το αποτέλεσμα και για τους καταναλωτές. 32% είναι πολύ καλό αποτέλεσμα. Ξεκινήσαμε στο 27, από το 27%, φτάσαμε το 32% και η πορεία μας είναι πάντα ανωδική. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο, περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ευχαριστώ, Σον. Ευχαριστούμε τον σκιώδη συγγητή μας. Άλλο σκιώδη συγγητής είναι ο συνάδελφος Τούρμες. Πραγματικά δείξαμε το καλύτερο πρόσωπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Καταπληκτικό ηγέτη, αλλά και ένα επιτελείο σχεδόν εισηγητών που πραγματικά ήταν ε, σύσσωμο. Ε, κάναμε μια συσπηρωμένη ομάδα και καταφέραμε από το 27% να πάμε στο 32% παρά την αντίθεση πολλών κυβερνήσεων και τα καταφέραμε. Μπράβο μας. Έχουμε την πανέμορφη ρήτρα αναθεώρηση επίσης που ε, δίνει μια σαφή μια τη ανωδική πορεία. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη. Στην πράξη σημαίνει ότι από την αρχική πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είχαμε 45% ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι το 2030, τώρα θα πάμε στο 60% και, και κάτι παραπάνω. 60 και, 60 και παραπάνω, αιωλική ενέργεια, υδροελεκτρική, ε, ηλιακή, βιομάζα, βιοενέργεια στην ηλεκτρική ενέργεια. Οπότε πολύ λιγότερο άνθρακα, ορυκτά καύσιμα και πυρηνική ενέργεια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Πραγματικά ήταν συντριπτική η επιτυχία και η νίκη μας. Και θυμάστε πριν από μερικού μήνες που στη Μαδρίτη σας είχα πει στο τέλος συνεδρίασης θα νικήσουμε Βενσερέμος και τα καταφέραμε. Ε. Χαίρομαι ιδιαίτερος. Ευχαριστώ κύριε Νίμπλερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ καλή δουλειά ε, και για την ε, πραγματικά δυναμική υποστήριξη των ε, θέσεων του Κοινοβουλίου και ευχαριστώ και τον πρόεδρο, ο οποίο ε, και αυτό στήριξε όλο αυτό τον μαραθών διαπραγματεύσεων. Ένα θέμα, κύριε Μπλανκολόπε, θέλω να πω. Αναφερθήκατε στο τέλο ε, στην ίδια κατανάλωση. Ε, γνωρίζω, μάλλον δεν γνωρίζω ακόμα τον συμβασμό στην τελική του εκδοχή. Είπατε ότι η ίδια κατανάλωση θα πρέπει να εξαιρείται φόρων και εισφορών αλλά εγώ το μόνο που θέλω να πω είναι να επισημάνω ότι για τη δική μας τη χώρα, όπου η ε, ήταν ήδη πολύ νωρίς, αυτό δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε υπερβολική στήριξη των μικρών εγκαταστάσεων. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα είδος ευελιξίας. Υπάρχει αυτή η ευελιξία στο συμβιβασμό, γιατί ξέρετε σε τελική ανάλυση οι πολλές εξαιρέσεις οδηγούν στο να πρέπει να καταβάλουν όλοι οι άλλοι πολίτες ε, το ποσό το οποίο προβλέπεται ως εισφορά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και Αγαπητοί φίλοι, συγχαρητήρια στον εισηγητή, πάρα πολύ καλή δουλειά, το είπαν αυτό και οι σκιώδεις μας και σας στηρίζω ανεπιφύλακτα. Εντυπωσιακό το αποτέλεσμα πολύ καλές διαπραγματεύσεις, δεν ήταν εύκολα όλα αυτά, αλλά βεβαίως ε, το Συμβούλιο ως συνήθως ε, εκπροσωπεί μια λιγάκι διαφορετική άποψη. Αλλά αυτή είναι η Ευρωπαϊκή μας Ένωση που σε γενικές ε, γραμμές νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε μια λύση, μπορούμε να είμαστε υπομονετικοί με πνεύμα συνεργασία στην Επιτροπή μας. Ευχαριστώ όλους τους και οδησηγητές και τον εισηγητή και τώρα πάμε όχι στο τελευταίο, αλλά αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε στη διάθεσή μας ακριβώς έξι λεπτά. Θα περάσουμε, μισό λεπτό λέει ο Πρόεδρος, έχουμε και την ενημέρωση της ε, αποστολής της Ήτρε στο Silicon Valley. Έχουμε ε, την διαχείριση της Ενεργειακής Ένωσης, έχουμε και τον Τούρμες και την κυρία Ρίβαση. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω όλους και οδησηγητές γιατί αν καταλήγουμε σε θετικά αποτελέσματα αυτό είναι χάρη στη συσπηρωμένη ομάδα που συστήσαμε και φυσικά στη συνεργασία με τον πρόεδρο. Ε, έτσι εξασφαλίσαμε την καλύτερη δυνατή διαχείριση και είχαμε σημαντική πρόοδο στον τρίτο άτυπο διά, τριμερή διάλογο. Και καταλήξαμε συμφωνία για το άρθρο 35 με τη Βουλγαρική Προεδρία θα έχουμε δύο επιτροπές, μία επιτροπή για, την, για τις κλιματικές αλλαγές και μία επιτροπή για την Ενεργειακή Ένωση, με σαφείς και ξεκάθαρες αρμοδιότητες για την κάθε επιτροπή. Επίσης, ε, η Ενεργειακή Ένωση θα επιληφθεί και τον οριζόντιο θεμάτων, η σχετική επιτροπή δηλαδή. Γιατί έχουμε την οδηγία για τις ανανεώσιμες πήγες ενέργειας, αλλά θέλουμε μια γενικότερη επιτροπή που θα εξασφαλίζει την ε, έμπρακτη εφαρμογή όλων των στόχων. Επίση, ε, συμφωνήσαμε επί τη αρχή για τη διάσταση τη ενεργειακή ασφάλεια, τη εσωτερική αγορά ενέργεια και τη ενεργειακή ένδυα. Επίση, συζητήσαμε και τις, ε, τη σχέση μεταξύ τη διαφοροποίηση τη προμήθεια στην ενέργεια, τη ανεξάρτητοποίηση από τι ε, εισαγωγέ και το δυναμικό της ενεργειακής αγοράς. Επίσης, ε, έχουμε κάποιες ε, τεχνικές ε, διατυπώσεις για τη δημιουργία των πάγιων και ελεύθερων τιμών, τις, τους μηχανισμούς ικανότητας και τις ζώνες προσφοράς. Για το μεθάνιο που έγινε, είχαμε μεγάλη διένεξη, τελικά καταλήξαμε σε ξεχωριστή παράγραφο 14α για το μεθάνιο. Η Βουλγαρική Προεδρία δέχτηκε την πρότασή μας να έχουμε ένα ευρωπαϊκό στρατηγικό σχέδιο για το μεθάνιο ε, και εμείς προσφέραμε κάποια ελαστικότητα σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια της προγραμματισμένης χρηματοδότησης για τις κλιματικές αλλαγές. Σε ό,τι αφορά τα τεχνικά θέματα, θα ήθελα να τονίσω ότι στηρίζουμε απόλυτα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα θέματα αυτά και θα πρέπει τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση να επιδείξουν διαφάνεια στην προγραμματισμένη χρηματοδότηση των κλιματικών αλλαγών των αναπτυσσόμενων χωρών. Γιατί έτσι θα βοηθήσουμε αυτέ τι αναπτυσσόμενε χώρε ε, για καλύτερο σχεδιασμό και πρόβλεψη. Επίση, ε, συμφωνήσαμε επί τη αρχή για την περιφερειακή συνεργασία και την μακροπεριφερειακή συνεργασία. Τελικά, η οριστικοποίηση του κειμένου θα γίνει σε τεχνικό επίπεδο. Έχουμε και ένα τέταρτο και ελπίζω τελευταίο τριμερή διάλογο που θα γίνει σήμερα το βράδυ και εκεί θα επιλύσουμε τα εκρεμή πολιτικά θέματα όπως τις πηγές τα, της ανανεώσιμης ενέργειας, το gap filler, το, το, την ενεργειακή απόδοση, τα εθνικά σχέδια και την ημερομηνία υποβολή των σχεδίων και της τελικής έγκρισης, καλώς και το χρονοδιάγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οπότε ε, έχουμε πολλά θέματα στην ημερήσια διάταξη για τον τελευταίο τριμερή διάλογο και θα, προσπαθούμε να το θα προσπαθήσουμε να τα ομαδοποιήσουμε ώστε να τα διεκπαιρεώσουμε όλα με στη νύχτα. Ελπίζω να είναι ο τελευταίος ε, τριμερής διάλογος ο σημερινός και να, τον, να βάλουμε την υπογραφή μας. Ελπίζω όχι ε, άγρια χαράματα, αλλά και κάπως νωρίτερα αν, καταφέ, τα καταφέρουμε. Οπότε θα έχουμε ένα Big Bang στις 7 το απόγευμα. Ε, Παράλληλα έχουμε και την ε, διάσκεψη των Πρόεδρων Επιτροπών. Θα κάνω ό,τι μπορώ. Ναι. Θα προσπαθήσω να είμαι πανταχού παρόν. Άλλη δυνατότητα δεν έχουμε γιατί έχουμε και τη σύγκρουση αρμοδιοτήτων στη διάσκεψη Πρόεδρων Επιτροπών. Αλλά θα δώσω το παρόν στον τριμερή διάλογο στις 7. Θέλετε να προσθέσετε κάτι κύριε Τουρμές. Νομίζω ότι έχουμε καλά προετοιμαστεί για τον τριμερή διάλογο του απογεύματος και έχουμε και εδώ μια πολύ αξιόλογη ομάδα και μια πολύ καλή συνεργασία μεταξύ των πολιτικών ομάδων, οπότε ε, έχω μεγάλη αισιοδοξία για το αποτέλεσμα. Τέλεια, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τους δύο συγητές και τους κοιόντες συγητές, γιατί είναι πολύ σημαντικό το θέμα της διακυβέρνησης της Ενεργειακής Ένωσης. Πολύ σημαντικό και για μας και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θερμά ευχαριστώ. Παρακαλώ, Ευχαριστώ, Γιέζη. Θα ήθελα να δώσω τα εύσημα στον Κλώτη Μισελ και τους και οδησυγητές των πολιτικών ομάδων και ευχαριστούμε και σε εσά. Εμείς θα ξεκινήσουμε στις 8, ελπίζουμε η ενεργειακή απόδοση να ολοκληρωθεί στις 7. Φυσικά πρώτα η ενεργειακή απόδοση, ε, ενεργειακή μετάβαση, καταπολέμηση ενεργειακής φτώχειας, και φυσικά διαβούλευση από τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Το είχε πει, Γέζη. Θέλουμε καθαρή ενέργεια για όλου του Ευρωπαίου πολίτε. Γιατί θα πρέπει να βάλουμε τον πολίτη στο επίκεντρο τη προσπάθειά μα. Επίση, χαίρομαι για το αποτέλεσμα που είχαμε στι ΑΠΕ. Και συγχαρητήρια στο Λόπε, στο Σον Κέλλη. Μπράβο σα. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ, αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι. Και φτάσαμε στο τελευταίο θέμα πριν τις τη μεσημβρινή διακοπή. Αποστολή της Ίντρε, της στην Silicon Valley. Ο κύριος Νίκα ε, είναι ο, ήταν επικεφαλής. Θα μας ενημερώσει όμως τα αγγλικά, γιατί σε ένα λεπτό θα διακοπεί η διερμηνία. Αλλά νομίζω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε στα αγγλικά. Ντάνι, είσαι έτοιμος? been seven members of the ITRE committee, together with our secretariat and